Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ήδη ένα τέταρτο καθυστέρηση. Καλό θα ήταν να αρχίσουμε. Θα ήθελα να ε, σας καλημερίσω όλους. Το πρώτο θέμα είναι η έγκριση της ημερήσης διάταξης. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μεταδίδεται στο διαδίκτυο οι συνεδρίες και ως συνήθως ε, οι ώρες που έχουμε προβλέψει στην ημερήσια διάταξη είναι ενδεικτικές. Ε, παρακαλώ να έρχεστε εγκαίρως στην συνεδρίαση για το θέμα σας. Δεν προτείνει κανείς ε, αλλαγή στην ημερήσια διάταξη και θα παρακαλούσα να την εγκρίνουμε χωρίς τροποποίησεις. Ωραία. Δεύτερον, ανακοινώσεις της Προέδρου. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ενδέχεται η συνεδρίαση των συντονιστών να ματαιωθεί, θα το δούμε αυτό κατά τη διάρκεια τη ημέρα θα το αποφασίσουμε. Ε, σχετικά με τις αποφάσεις προηγούμενης συνεδρία συντονιστών, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ελήφθη απόφαση για τις νομοθετικές εκθέσεις σχετικά με τον ειδικό φόρο κατανάλωση στη Μαδέρα και τις Ασόρες να επεκταθεί ο μειωμένος συντελεστής. Ε, εκεί θα επιλέξουμε την απλουστευμένη διαδικασία που σημαίνει ότι η πρόεδρος της Επιτροπής ε, θα κάνει τη σχετική γνωμοδότηση, είναι δικό της καθήκον και σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού θα εγκριθεί αυτό, δηλαδή χωρίς και τροπολογίες. Είναι το σημείο 6 σήμερα στην ημερήσια διάταξη για την μη νομοθετική γνωμοδότηση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, τον τρόπο που έγιναν διαπραγματεύσει, τι διδάγματα πρέπει να εξαγάγουμε για το μέλλον. Το ΕΛΚ πήρε την έκθεση, η συγγητής είναι ο κύριος Όλμπριχτ. Ε, είναι στην Επιτροπή Προϋπολογισμών η έκθεση, εμείς κάνουμε γνωμοδότηση. Ε, ε, θα το συζητήσουμε σήμερα. Επίσης, οι συντονιστές αποφάσισαν να συστήσουν ακύρωση των ημερών συνεδριάσεων, οι υπόλοιπε συνεδριάσει μας δηλαδή να γίνονται σε μία μέρα. Σήμερα έχουμε πιο σύντομη συνεδρίαση, ε, μία ημέρας, όχι δύο ημερών πλέον και η επόμενη συνεδρίαση πότε έχει προβλεφθεί 19 και 20 Μαρτίου, δεν θα είναι διήμερη, θα περιοριστεί σε μία ημέρα στις 19 του μηνός. 19 Μαρτίου η επόμενη συνεδρίαση και θα προσπαθήσουμε το απόγευμα να ψηφίζουμε κιόλα. Δηλαδή περιορίζεται η διάρκεια των συνεδριάσεων που μας απομένουν. Αυτά αποφάσισαν οι συντονίστες. Θα προχωρήσουμε στο σημείο 3 στην ημερήσια διάταξη που είναι η συζήτηση της εξωτερικής μελέτης η οποία ε, είχε παραγγελθεί από την Επιτροπή μας και εφαρμόστηκε από τη Διεύθυνση για ε, Διαρθρωτικές Πολιτικές εξωτερική μελέτη σχετικά με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση και την Πολιτική Συνοχή. Έχουμε δύο ε, ερευνητές που εργάστηκαν στη μελέτη αυτή, τον κύριο Ιαν Μπέκ, ε, καθηγητή στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο του London School of Economics and Political Science. Έχουμε και τον Τζον Μπάχτελ από το Πανεπιστήμιο Strathclyde της Γλασκόβης. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση θα ήθελα να σας δώσω το λόγο με τη σειρά που εσείς αποφασίσετε για να παρουσιάσετε τη μελέτη. Ο Μπέκ θα ξεκινήσει. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για τη δυνατότητα που μας δίνετε να παρουσιάσουμε τη μελέτη αυτή και θα προσπαθήσουμε να αναφερθούμε σε κάποια από τα σημαντικότερα σημεία της έκθεσής μας αυτής τα 20 λεπτά που μας δίνεται εν είδη εισαγωγής. Ίσως να με βοηθήσει κάποιος από το τεχνικό προσωπικό για να μπορέσω να προβάλλω την παρουσίασή μου. Καταρχάς πρέπει να πούμε Περιμένουμε να καθαρίσει πρώτα η οθόνη. Μπορεί κάποιος να βοηθήσει τον... Μάλλον λειτουργεί πλέον, ωραία. Ασχοληθήκαμε λίγο με την φύση των μεταρρυθμίσεων οικονομικής διακυβέρνησης και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι έχουμε τέσσερις βασικές κατηγορίες μεταρρυθμίσεων. Η πρώτη κατηγορία, όπως βλέπετε εδώ, είναι η νομισματική πολιτική. Έχουν γίνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της νομισματικής πολιτικής όπου βλέπουμε μία επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μπορούμε να πούμε πλέον ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει γίνει ένας παράγοντας, τύχη κάπως μπορούμε να πούμε, στην πολιτική συνοχή. Και αυτό γιατί οι δράσεις πλέον της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση που κάνουμε. Πώς συμβαίνει τώρα αυτό στην πράξη βλέπουμε ότι εμέσως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γίνεται ο δανειστής σε εσχάτη ανάγκη μπορούμε να πούμε. Πάλι κάτι δεν λειτουργεί καλά. Και έτσι λοιπόν η δανειοδότηση αυτή σε έσχατη ανάγκη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γίνεται όταν αυτή αγοράζει ομόλογα στην δευτερεύουσα αγορά και κατά αυτόν τον τρόπο μειώνεται το κόστος χρηματοδότησης για τις χώρες εκείνες οι οποίες έχουν πετύχει το χαμηλότερο αυτό κόστος. Επίσης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει σημαντικότατο ρόλο στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Αυτές είναι οι σημαντικότερες αλλαγές που έχουμε στην πρώτη κατηγορία μεταρρυθμίσεων στον τομέα της νομισματικής πολιτικής. Περνάμε σε μια δεύτερη κατηγορία στο Fiscal Compact, το Δημοσιονομικό Σύμφωνο και σε όλες τις άλλες αποφάσεις που επηρεάζουν τελικά την πολιτική εποπτείας και επιθαρχίας των κρατών μελών. Ουσιαστικά αναφερόμαστε όλο και περισσότερο στην χρηματοπιστωτική πειθαρχία, αλλά ξέρετε ότι η διαδικασία μακροοικονομικής ανισορροπίας και κυρίως ο σχετικός συντονισμός πλέον των κρατών μελών επηρεάζουν έντονα τις μακροοικονομικές πολιτικές και έχουν επιπτώσεις σε διάφορα προβλήματα, όπως για παράδειγμα σε προβλήματα στον ε, κρατικό ισολογισμό ή σε προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν πολλές φορές με, τη με την φούσκα που προκαλείται στα ακίνητα. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά μετατρέπεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς επίσης και άλλων παραγόντων στο ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τις αποφάσεις των κρατών μελών για τη μακροοικονομική πολιτική. Η επόμενη κατηγορία μεταρρυθμίσεων είναι ρυθμιστικής φύσης βλέπουμε ότι υπάρχουν νέες μορφές εποπτείας, παρακολούθησης, μακροπροληπτικής εποπτείας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, για παράδειγμα, και έχουμε και κάποιες αλλαγές οι οποίες επέρχονται όλο και περισσότερο στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία γίνεται πλέον υπεύθυνη για τον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας. Και περνάμε κατά αυτόν τον τρόπο στην τέταρτη κατηγορία μεταρρυθμίσεων, όπου ουσιαστικά βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και κυρίω η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχουν νέε αρμοδιότητε επί των κρατών μελών. Και κατά αυτόν τον τρόπο τροποποιεί τη δημοκρατική ισορροπία για το ποιο κάνει ακριβώ τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιε είναι οι άμεσε επιπτώσει όλων αυτών. Βλέπουμε ότι ο βασικός ρόλος για την οικονομική διακυβέρνηση έγκυται πλέον στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Έχουμε χάσει κάποιες άλλες διαδικασίες οι οποίες είναι λιγότερο ορατές, όπως για παράδειγμα η Ευρώπη 2020. Δεν ακούμε όμως πάρα πολύ συχνά πλέον για την πολιτική αυτή. Ακούμε όλο και περισσότερο για πολιτικές που συνδέονται με το ευρωπαϊκό εξάμεινο και ακούμε όλο και λιγότερο για τις ε, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ε, στρατηγικές του προγράμματος Ευρώπη 2020. Ο συντονισμός επίσης αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο του νέου αυτού συστήματος. Υπάρχουν πάρα πολλές αποφάσεις που λαμβάνονται πλέον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και που απαιτούν καλύτερο συντονισμό των κρατών μελών πλέον. Δεν τυχαίο ότι η διακυβερνητική ε, συνθήκη ονομάζεται πλέον συνθήκη συντονισμού. Και βέβαια δεν γνωρίζουμε σε ποιο σημείο μπορούμε να φτάσουμε με το συντονισμό, αν υπάρχουν όρια στο συντονισμό αυτό. Και βέβαια έχουμε και επιπτώσεις στην πολιτική συνοχή στη συνέχεια. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου επίσης είδαμε ότι ήταν 27 τα κράτη-μέλη τα οποία ήταν εναντίον ενός μόνο κράτους μέλους της Γερμανίας και είχαν και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την υποστήριξη του Herman Van Rompuy, καθώς προσπαθούσαν να προωθήσουν όλο και περισσότερο τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών. Υπήρχαν, υπήρχαν κράτη-μέλη τα οποία δεν ήθελαν κάτι τέτοιο και επιθυμούσαν να υπάρχουν λιγότεροι, μια μικρότερη σύναψη συμβάσεων όσον αφορά την πολιτική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, έχουμε ακούσει και πολιτικούς ηθήνοντες όπως ο Φρανσουά Αλόντ, ο οποίος ε, κατέκρινε τις αποφάσεις αυτές που έχουν ληφθεί τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την πολιτική συνοχή και τη γενικότερη τάση προς μία όλο και υψηλότερη, μεγαλύτερη μάλλον σύναψη συμβάσεων βλέπουμε ότι στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής συνάπτονται πλέον συμβάσεις ανάμεσα στο κράτος μέλος ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή μια περιφέρεια και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία δεν δέχονται την προσέγγιση αυτή. Μας λένε ότι αυτό το οποίο αρχικά ονομάζαμε CCI, δηλαδή μέσω ανταγωνιστικότητας και σύγκλησης, ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο επινόησε η γερμανική κυβέρνηση και με το οποίο αντιτίθενται τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Είναι αβέβαιο λοιπόν μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να φτάσουμε με το συντονισμό. Κάτι το οποίο επίση είναι αβέβαιο είναι ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλο αυτό το σύστημα. Θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιβλέπει τελικά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στι νέε αρμοδιότητέ τη. Θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβλέπει επίση και το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλέ αντιπαραθέσει αυτή τη στιγμή, οι οποίε πρέπει να επιληθούν. Ποιε είναι οι βασικέ τώρα επιπτώσει. Στα πλαίσια της χάραξης πολιτικής βλέπουμε κυρίως ότι οι εθνικοί προπολογισμοί όλο και περισσότερο θα περιορίζονται, θα ασκείται πίεση σε αυτούς και θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επίβλεψη και εποπτεία από ό,τι στο παρελθόν. Και αυτό το βλέπουμε ιδίως στις χώρες εκείνες οι οποίες έχουν αντιμετωπίσει τις ε, περισσότερες δυσκολίες στο παρελθόν. Να φέρουμε μόνο στις χώρες εκείνες οι οποίες υπάγονται σε μνημόνια κατανόησης δημοσιονομικής προσαρμογής. Αναφέρομαι ακόμα και σε χώρε όπως η Ισπανία και η Ιταλία που έχουν αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα με τους εθνικούς προπολογισμούς τους και το ίδιο ισχύει ακόμα και για τον Ηνωμένο Βασίλειο, στο οποίο έχουν ληφθεί μέτρα λιτότητος. Ο τρόπος λοιπόν που δαπανούνται πλέον τα δημόσια χρήματα, οι δημόσια πόροι θα τροποποιηθεί. Θα ασκείται δηλαδή στι δημόσιε αυτέ δαπάνε όλο και μεγαλύτερη εποπτεία και τελικά πίεση. Και αυτό προφανώ θα πειράσει τι επενδύσει και κυρίω τι δημόσιε επενδύσει που γίνονται στα κράτη-μέλη και οι οποίε συνδέονται με την πολιτική συνοχή. Αυτό σημαίνει κατ' επέκταση ότι οτιδήποτε μπορεί να δαπανηθεί σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο θα επηρεάζεται όλο και περισσότερο από αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα μας απασχολεί όλο και περισσότερο η ποιότητα των επενδύσεων αυτών, αν πραγματικά μπορούν να οδηγήσουν σε οικονομική ανάπτυξη. Ξέρετε βέβαια ότι αν καταφέρουν οι οικονομολόγοι να, βρούνε το, να λύσουν το μυστικό αυτό, να καταφέρουν να μας πούνε πώς μπορούμε να πετύχουμε οικονομική ανάπτυξη εύκολα, θα γινόμασταν όλοι πολύ εύκολα πλούσιοι. Επίσης βλέπουμε όλο και περισσότερο ότι η πολιτική συνοχή συνδέεται όλο και περισσότερο με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 και αυτό το δούμε όλο και περισσότερο στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Αν εξετάσουμε λοιπόν τώρα το σύνολο του νέου αυτού συστήματος, βλέπουμε ακόμα ότι υπάρχουν προβλήματα και αδυναμίες. Θα ασχοληθώ με το ζήτημα αυτό λίγο αργότερα. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει ακόμα επιληθεί. Η τοξική αυτή σχέση επιφύσταται ακόμα μεταξύ των τραπεζών και της χρηματοδότησης των κρατών μελών, του δημοσίου χρέους δηλαδή που έχουμε στα κράτη-μέλη. Το ζήτημα αυτό δεν έχει ακόμα επιληθεί και θα έχουμε βέβαια και νέε επιπτώσεις εξαιτία των νέων αυτών μεταρρυθμίσεων που ανέφερα. Επίση, η Τραπεζική Ένωση δεν έχει επιλύσει όλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Υπάρχουν κάποια όρια και περιορισμοί αυτή τη στιγμή στις αρμοδιότητε τη Τραπεζικής Ένωση, ιδίω όσον αφορά τι τελευταίε αποφάσει που ελήφθησαν για τον νέο μηχανισμό εξυγίανση. Και ξέρετε ότι με τις πρόσφατες αποφάσεις γερμανικού δικαστηρίου βλέπουμε ότι ασκείται όλο και μεγαλύτερη πίεση από τα κράτη-μέλη, εν προκειμένου από τη Γερμανία και από την Bundestag, που δεν επιτρέπουν πλέον στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν ελεύθερα τους πόρους τους στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής. Και βλέπουμε λοιπόν ότι γεννιούνται όλο και νέες διαδικασίες που επηρεάζουν προφανώς όλο το σύστημα δημοσίων δαπανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δώσω τώρα το λόγο στον αδελφό μου. Thank you, um, Ευχαριστώ, Ιαν. Καλημέρα σας, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Να περάσουμε στις συνέπειες της οικονομικής διακυβέρνησης στην πολιτική συνοχή. Στη μελέτη θέσαμε στους αυτούς μας τέσσερας, τέσσερις ομάδες ερωτήσεων. Η πρώτη είναι πως η πολιτική συνοχής συνεισφέρει στην οικονομική διακυβέρνηση. Έπειτα ποιε είναι οι συνέπειες των κατευθύνσεων που παίρνει η οικονομική διακυβέρνηση για την πολιτική συνοχής. Τρίτον, δεδομένων των προσανατολισμών αυτών που είναι κάπως αβέβαιοι, τι είδους σενάρια θα μπορούσαμε να επινοήσουμε για τι σχέσει μεταξύ οικονομική διακυβέρνηση και πολιτική συνοχή και τέλο ποιε είναι οι συνέπειε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση, την ε, συμβολή της πολιτικής συνοχής στην οικονομική διακυβέρνηση. Προφανώς η πολιτική συνοχής ε, έχει σκοπό να ενδυναμώσει ε, την σύνοχη την ίδια, αλλά πρέπει να συνεισφέρει και στη μακροοικονομική διακυβέρνηση με διάφορους τρόπους. Ε, ή τουλάχιστον αυτό συμβαίνει στην πράξη. Υπάρχει η λειτουργία της συμμόρφωσης με τους μακροοικονομικούς κανόνες, κάτι που εδώ και 20 χρόνια υπήρχε σε σχέση και εξαιτία του Ταμείου Συνοχής, με ένα ιστορικό όμως αρκετά ανάμεικτο, δηλαδή κάποια κράτη-μέλη να συμμερφώνονται με την αιρεσιμότητα ενώ κάποια άλλα όχι οπότε πρόσφατα να έχουν και αναστολή της χρηματοδότησής τους. Όμως ακούστηκε ότι είναι πλέον πιο ξεκάθαρα τα δείγματα που πρέπει να ακολουθηθούν και ότι υπάρχει και η απειλή του επονιδισμού ε, για αυτούς που δεν συμμορφώνονται. Πάντως η αιρεσιμότητα έχει επεκταθεί σε όλα τα διευθυντικά και επενδυτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια ε, ε, υγιέστερη οικονομική διακυβέρνηση, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με τις συστάσεις του Συμβουλίου και το καθεξής. Υπάρχει περιθώριο για ανάληψη δράσης ως προς τις συμφωνίες εταιρική σχέσης, τα λειτουργικά προγράμματα και βεβαίως ακριβώς επειδή υπάρχει και η δυνατότητα αναστολής των πληρωμών. Θα μιλήσω για τις συνέπειε, θα δώσω λίγο. Έπειτα, η πολιτική συνοχή έχει μια λειτουργία σταθεροποίηση, ιδίω κατά την περίοδο τη κρίση. Έχει ενισχύσει την ανάκαμψη σε πολλέ περιπτώσει και αυτό έχει διαπιστωθεί στην πράξη. Έχουμε δει επαναπρογραμματισμό σε κάποιες χώρες με την δυνατότησή του και τι δαπάνε, όπω με τη δημιουργία θέσεων απασχόληση και τι επενδύσει, ενώ σε κάποιες άλλες ο επαναπρογραμματισμός που έχει προκληθεί από τον προγραμματισμό της πολιτικής συνοχής έχει μεταφέρει την ε, έμφαση των, των προγραμμάτων σε μακροπρόθεσμους και περιφερειακούς στόχους. Κατά τρίτον, η πολιτική συνοχής όλο ένα και περισσότερο συντελεί στη ε, δημιουργία, στην ανάπτυξη την ίδια και τις περισσότερες δαπάνες σε ορισμένους τομείς. Είδαμε το τελευταίο διάστημα με τη στατικική της Λισαβόνας και τις απαιτήσει εντοπισμού κονδυλίων, μετατόπιση των δαπανών της πολιτικής συνοχής προς ε, συγκεκριμένες κατηγορίες όπως η έρευνα και η καινοτομία. Υπήρξε δηλαδή σημαντική αύξηση στην αναλογία των δαπανών που αποδόθηκαν, που κατευθύνθηκαν σε αυτούς τους συγκεκριμένους τομείς υπό την στρατηγική της Λισαβόνας. Αυτό με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο βλέπουμε να εντείνεται, καθώς και με την ε, επικέντρωσή μας στην Ευρώπη για το 2020. Υπάρχει όμως και αυξανόμενη ε, επικέντρωση σε τομείς, σε συγκεκριμένους τομείς των δαπανών. Τομεακή προσέγγιση και πολλαπλές προϋποθέσεις που πολλές φορές είναι και αντικρουόμενες αντιφατικέ μεταξύ του. Τέλο, η πολιτική συνοχή διδραματίζει και ένα συγκεκριμένο ρόλο στο να ενισχύει, να εισάγει την τοπική, την εδαφική διάσταση των δαπανών προκειμένου να ανταποκριθεί σε υποεθνικές ανάγκες και προκλήσεις αλλά και από το πολυεπίπεδο μοντέλο διακυβέρνησης αναγκάζεται να εμπλέξει τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης την λήψη αποφάσεων και την κατανομή των πόρων. Επίσης υπάρχει και μια λειτουργία συντονισμού ή τουλάχιστον η δυνατότητα συντονισμού ε, τομέων πολιτικής, χάραξης πολιτικής και καθορισμό κοινών στόχων. Το ερώτημα ποιες είναι οι συνέπειες από τις μεταρρυθμίσεις στην οικονομική διακυβέρνηση για τη χάραξη πολιτικής. Το σημείο αφετηρίας είναι η υγιής, είναι το να υπάρχει ένα υγιές και σταθερό και αξιόπιστο οικονομικό περιβάλλον και αυτό επιτρέπει τις επενδύσεις διότι ε, ε, τα επιτόκια και η διακύμανση των τιμών και οι διαρκείς μεταβολές ε, αυξάνουν την απόσταση μεταξύ φτωχών και πλουσίων στις περισσότερες περιοχές. Αλλά εδώ υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να υπογραμμίσουμε. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ της σοβαρής πίεσης στα δημοσιονομικά με δημοσιονομικές και διαφθορτικές μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν τον προγραμματισμό των δημοσιονομικών κάθε κράτους με μακροπρόθεσμες συνέπειες. Υπάρχουν εδώ περισσότερες περικοπές, ε, περιορισμοί και περικοπές στην ε, στα κονδύλια που αφορούν την ανάπτυξη. Αυτό περιορίζει και τα, τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής. Και αυτό ανησυχεί ιδιαίτερο σε χώρες όπως η Ελλάδα ή η Πορτογαλία σε αυτή τη φάση. Εκεί όπου η πολιτική συνοχής είναι το μεγαλύτερο, εάν όχι ολόκληρο το κομμάτι της ε, χρηματοδότησης. Βλέπετε λοιπόν αντιφατικούς στόχους στην πολιτική συνοχή. Αλλά υπάρχουν και συνέπειες από τις προϋποθέσεις που προκαλούνται από τις μεταρρυθμίσεις στην οικονομική διακυβέρνηση, όπως αυτές θα πρέπει να εφαρμοστούν στην χάραξη πολιτικής. Ανέφερα τις διατάξεις που έχουν να κάνουν με τον, με τον επαναπρογραμματισμό και την κατανομή των δαπανών. Το θέμα είναι πόσο εφικτές και αξιόπιστες είναι αυτές οι αλλαγές κάποιες φορές είναι δυσνόητες και όχι τελείως σαφείς. Υπάρχουν ε, προσεγγίσεις που είναι αρκετά τεχνοκρατικές από πάνω προς τα κάτω και είναι δύσκολο να ε, διακρίνει κανείς ποιο είναι το καλύτερο συμφέρον, το συμφέρον ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους. Και υπάρχουν και κάποια κράτη τα οποία ουσιαστικά γνωρίζουν συνέπειες που δεν μπορούν να καλύψουν ενώ άλλοι δικαιούχοι, περιοχές, περιφέρειες, τμήματα της κοινωνίας που δεν αναλαμβάνουν ευθύνη για προβλήματα τα οποία οδήγησαν συνολικά στις αλλαγές της μακροοικονομικής πολιτικής. Κατά τρίτον, όπως είπα και προηγουμένως, βλέπουμε να υπάρχει μεγαλύτερη έμφαση στους ε, στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως με την Ευρώπη του 2020 και βλέπουμε η πολιτική να ακολουθεί την κατεύθυνση των διευθυντικών μεταρρυθμίσεων και της χρήσης των παρεμβάσεων της πολιτικής συνοχής καθώς και τη στήριξη της διορθωτικής πολιτικής και των στόχων της ως συμπλήρωμα. Υπάρχουν αντιφάσεις βέβαια και εδώ Ω προ τους στόχους ενοχής κυρίω αλλά και στην πράξη, το θέμα είναι αν η πολιτική είναι σε θέση να επιτύχει τους στόχους αυτούς. Είδαμε ήδη τι δυσχέρειες αντιμετώπισαν τα κράτη-μέλη για να διαπραγματευτούν με τις υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής την συμμόρφωση με τις προσδοκίες τους ως προ του θεματικού στόχου και τι απαιτήσει για μεγαλύτερη ευελιξία Επίσης, ως προς την Τραπεζική Ένωση υπάρχουν εδώ ενδεχόμενα ωφέλη όπως καλύτερες και πιο ομοιόμορφες συνθήκες χρηματοδότησης, όριμα χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Οπότε έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί ο κατακαιρματισμός των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Και υπάρχουν και θεσμικές συνέπειες, κυρίως ως προς την ενδυνάμωση του ρόλου του Συμβουλίου, γιατί θα είναι το κέντρο της ε, λήψη στρατηγικών αποφάσεων, αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως προς τον εκτελεστικό της ρόλο. Θα παρακολουθεί δηλαδή τι συμφωνίε εταιρική σχέση και τα λειτουργικά προγράμματα. Οι συνέπειε για το Ευρωκοινοβούλιο είναι ακόμη κάπως ασαφεί, αλλά θα πω περισσότερα γι' αυτό εντό ολίγου. Τώρα να στραφούμε στα διαφορετικά σενάρια, στις υποθετικές καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν. Ε, συζητήσαμε σε δύο κεφάλαια τις υποθέσεις αυτές. Μία, αυτή που έχουμε ονομάσει την εκδοχή της περιορισμένης πραγματικής οικονομικής και νομισματικής ένωσης και δεύτερη, ε, δεύτερη υπόθεση την, ε, την, την πιο σφαιρική, την πιο ολοκληρωμένη ένωση. Στην ε, περιορισμένη εκδοχή έχουμε τις ήδη συμπεφωνημένες ε, αλλαγές στην κυβερνοτική πολιτική για την περίοδο από το 2013 και το 2014 έως 20. Τα βλέπετε και στην οθόνη πιο ξεκάθαρα, αλλά αναπτύσσονται και στη μελέτη με, το, με τη γραφική παράσταση της σελίδας 54. Ε, βλέπετε τα επίπεδα χρεών των κρατών μελών ως αναλογία του ΑΕΠ τους στον οριζόντιο άξονα και έπειτα στον κάθετο το πώς κατανέμονται τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής. Έτσι μπορούμε να έχουμε τέσσερις ομάδες χωρών, αυτές με υψηλά επίπεδα χρέους αλλά και μεγάλη έμφαση στις δαπάνες πολιτικής συνοχής, Κύπρος, Ελλάδα, ε, Ουγγαρία, Μάλτα και Πορτογαλία. Δεύτερον, χώρες με υψηλό χρέος αλλά χαμηλή χρηματοδότηση ε, της πολιτικής συνοχής, Αυστρία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τρίτον, χώρε χωρί χρέο, αλλά με μεγάλε δαπάνε στην πολιτική συνοχή. Πολλέ ήταν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 12 και έπειτα αυτέ με χαμηλή χρηματοδότηση ούτω ή άλλω, όπω η Δανία, η Σουηδία και η Φινλανδία κυρίως οι χώρες της πρώτης κατηγορίας έχουν τις μεγαλύτερες, δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις δημοσιονομικής προσαρμογής και βεβαίως εκεί υπάρχουν και καταστροφικότερες συνέπειες, ιδίως εάν υπάρξουν εθνικές, ε, μάλλον αναστολή των πληρωμών σε εθνικό επίπεδο λόγω μη συμμόρφωσης. Ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου σε αυτό το σενάριο, σε αυτή την εκδοχή, είναι να παρακολουθεί και να ελέγχει, αυξάνοντα το μέγιστο δυνατό βαθμό την ε, αρμοδιότητά του να παρακολουθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο και να δει κατά πόσον ε, υλοποιούνται υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές. Βεβαίως όλοι οι κανονισμοί αφήνουν μεγάλα περιθώρια γι' αυτό και το θέμα είναι πώς ερμηνεύονται όλα αυτά και στην πράξη. Όμως είναι σημαντικό από την άποψη της ε, δημόσιας λογοδοσίας. Τώρα, στο συνολικότερο σενάριο για την πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση σημαίνει ότι θα υπάρχει περισσότερο παρεσματισμό στα δημοσιονομικά των κρατών μελών με μια πραγματική τραπεζική ένωση και υπερεθνικά δημοσιονομικά μέσα για τη σταθεροποίηση και τους στόχους της. Εδώ οι συνέπειες είναι τελείως αστάθμητες, όμως πιστεύουμε ότι μια τέτοια δημοσιονομική εξουσία μπορεί να υποβαθμίσει την πολιτική συνοχή με λιγότερη χρηματοδότηση, εκτός και αν αυξηθεί σημαντικά ο προπολογισμό, πράγμα που θα έχει συνέπειες για την εδαφική και θεματική κάλυψη που προσφέρει αυτή η πολιτική. Επίσης, Μπορεί να υπάρχουν παρεμβατικότερες προϋποθέσεις και όρες σε σχέση με τις προσφατότερες ε, μεταρρυθμίσεις, με ε, συνέχιση των τάσεων που είδαμε τα τελευταία χρόνια και την ε, επιβολή της αιρεσιμότητας με αυτόματες κυρώσεις, την πάυση προγραμμάτων αλλά και εντάσεις πολιτικές και διοικητικές και δημοσιονομικές όπως είδαμε στην πρόσφατη περίοδο. Μία τέτοια ένωση θα μπορούσε να προβλέψει και νέα εργαλεία εάν δεν έχουν ήδη σχεδιαστεί όπως με περισσότερη έμφαση στους συγκεκριμένους τομείς και την ε, διάλυση του μοντέλου χρηματοδότησης από τον προπολογισμό όπως το έχουμε δει ως τώρα. Πάντως, τα νέα εργαλεία μπορούν να τα αλλάξουν όλα και αυτό θα εξαρτηθεί και από το μέγεθο ε, του προπολογισμού που θα προβλέπετε. Ένα μικρό προπολογισμό μπορεί να έχει περιορισμένο αντίκτυπο, ένα όμω μεγαλύτερο προπολογισμό μπορεί να είναι ανταγωνιστικό, να φέρει ανταγωνισμό από άλλε πολιτικέ στην πολιτική συνοχή. Και μπορεί έτσι να υπάρχει περισσότερη έμφαση σε εδαφικά και θεματικά σημεία και στόχους. Βέβαια, θα μπορούσε να απελευθερωθεί η πολιτική συνοχή από τη λειτουργία σταθεροποίηση που έχει αναλάβει και να δίδεται μεγαλύτερη προσοχή στον τρόπο που υλοποιείται στην πράξη. Τέλος, ως προς τα ερωτήματα που θέσαμε και το ποιες είναι οι συνέπειες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιλέξαμε τέσσερα σημαντικά μηνύματα, ομάδες ε, επιπτώσεων. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται να αναλάβει ισχυρότερο ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον σχεδιασμό των λειτουργιών των μέτρων της πραγματικής ε, οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Αυτό όπως εφαρμόζεται ως σήμερα για το ρυθμιστικό πλαίσιο δεν έχει αφήσει πίσω το ένα καλό ιστορικό. Μπορεί όμως το Κοινοβούλιο να παρακολουθεί πώς τα υπάρχοντα μέσα υλοποιούνται και αυτό πραγματικά δείχνει ότι και στο μέλλον χρειαζόμαστε ένα ισχυρό κοινοβούλιο σε αυτή τη λειτουργία. Έπειτα και στο κοινοβούλιο συζητείται αυτό ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερο συντονισμό μεταξύ των επιτροπών και περισσότερο διάλογο. Δεν είναι λοιπόν θέματα αυτά μόνο τη Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων των Προπολογισμών. Η σημασία τη πολιτική ε, συνοχή, των διευθυντικών ταμείων, του Ταμείου Συνοχή, με το ρόλο που έχω ήδη υπογραμμίσει, απαιτούν καλύτερο συντονισμό όλων των κοινοβουλευτικών επιτροπών και των ε, υπηρεσιών τους. Τρίτον, νομίζω το Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρακολουθεί καλύτερα πώς τα μέτρα ε, της Νομισματικής και Οικονομικής Ένωσης επηρεάζουν τα κάτι μέλη. Ιδίως τα ισχύοντα μέτρα για το ερχόμενο χρονικό διάστημα, αλλά και για τον ενδεχόμενο αντίκτυπο από μελλοντικέ μεταρρυθμίσεις ανέφερα τις εντάσεις που προκαλεί η οικονομική διακυβέρνηση στην πολιτική συνοχή, το πώς αυτά θα επηρεάσουν τα επιμέρους κρατημέλη, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στις συγκεκριμένες περιφέρειες και επαρχίες στα κρατημέλη είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Και έπειτα για την εξωτερική ανάθεση της διακυβέρνησης, την επέκταση αυτή των ε, συμβάσεων διαρκώς και την μετατόπιση του κέντρου λήψης αποφάσεων εκτός του δημόσιου χώρου, Αυτά όλα ε, μας κάνουν να απαιτούμε ένα πιο ισχυρό κοινοβούλιο που να κάνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κάτι μέλη υπεύθυνα για να λογοδοτούν. Να ολοκληρώσω σύντομα προσπαθώντας να ανακεφαλαιώσω όσα είπαμε. Πρώτον λοιπόν, σημαντικές αλλαγές. Σημαντικές αλλαγές που θα αλλάξουν το τοπίο για τους ε, εθνικούς φορείς και διεθνώς και τοπικός και εξαιτίας βασικά της ε, ευρωπαϊκής χαράξης πολιτικής. Υπάρχει εμέσω πλην σαφώ ένα νέο ρόλο, ένα de facto ρόλο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που καθορίζει ε, έστω και συμπτωματικά στόχου για την πολιτική συνοχή. Και έπειτα σίγουρα θα συνεχίσουν να υπάρξουν πιέσει τη δανειοδότηση από τράπεζε. Είδαμε τον κατακαιρματισμό τη χρηματοδοτική αγορά στην Ευρώπη, το τι γίνεται με τι μικρέ επιχειρήσει και τη δυνατότητά του να ανακάμψουν. Δεύτερο σύνολο συμπερασμάτων δεν γνωρίζουμε πραγματικά τι θα γίνει με την πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση και τι κατεύθυνση θα πάρει. Ξέρουμε ότι η Τραπεζική Ένωση είναι μία ε, λύση που δεν ικανοποιεί. Για την ώρα δεν υπάρχουν άλλες προτάσεις να υπάρξει ένα κοινό ε, ταμείο εγγύησης των καταθέσεων ώστε να αποφύγουμε τις τοξικές συνέπειες της λειτουργίας των τραπεζών για τα κρατημέλη και υπάρχει ένας ε, κίνδυνο που ελοχεύει φέτο, διότι καθώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αναλάβει την εποπτεία με τι δοκιμασίε ε, αντοχή που θα διεξαγάγει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, αυτό μπορεί να σημαίνει και άλλα προβλήματα. Στα κράτη-μέλη της χώρες που θα υπάρξουν προβληματικές τράπεζες δεν θα είναι απλό να εξηγιανθούν ή να διασωθούν αυτές. Μπορεί λοιπόν να προκύψουν προβλήματα χρηματοδότησης. Οι προτάσεις για τη Δημοσιονομική Ένωση έτσι κι αλλιώς σε τέλμα παρά το γεγονός ότι ανακοινώθηκαν στο blueprint, στο αποτύπωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με συγκεκριμένους στόχους δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις ούτε για τις δυνατότητες δαπανών ούτε για τα ευρωομόλογα. Αν υπάρχουν Γερμανοί στην αίθουσα θα μας πούνε nein, Μόνο που θα ακούσουν τη λέξη ευρωομόλογα και οι Φιλανδοί φαντάζομαι. Ο κίνδυνος λοιπόν εδώ είναι οι φιλοδοξίες ε, της προβλεπόμενης αυτής ένωσης να μην ε, τελικά υλοποιηθούν ποτέ. Και τέλος αυτό που έχουμε τονίσει επανειλημμένως για την νομιμοποίηση των στόχων ε, της οικονομικής διακυβέρνησης και της πολιτικής συνοχής υπάρχουν πραγματικά ακόμη πολλές προκλήσεις. Πρόεδρος, ευχαριστούμε Ιαν, ευχαριστούμε Τζον. Η σιωπή ήταν φαντάζομαι δείγμα ότι σας ακούσαμε με προσοχή και μας επηρεάσατε στο πώς βλέπουμε το μέλλον. Να δώσω το λόγο στους συναδέλφους για ερωτήσεις και σχόλια. Είναι λίγοι εδώ παρόντες, αλλά έχετε το λόγο. Ε, ο Γιάνν πρώτος ή ο... Υπολφείτε μεταξύ σας ποιος θέλει πρώτος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σκεφτόμουν κάτι σχετικά με τη συμπληρωματικότητα. Πρόσφατα είχα την ε, τύχη να ακούσω, ξέρεις, τον Υπουργό κύριο Σόιμπλε, όταν παρουσίασε τις δικές του απόψεις για το μέλλον της οικονομικής διακυβέρνησης Ευρωζώνης και τα και το μελλοντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς επίσης και την ανάγκη να συσταθεί νέο κοινοβούλιο για τις χώρες Ευρωζώνης. μετά την ε, παραδοχή ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, και αν τον παραθέτω σωστά, δεν προσφέρονται ή δεν είναι σε θέση σύμφωνα με τη συνθήκη να διαχειριστούν τα προβλήματα της Ευρωζώνης. Άρα χρειάζεται αναθεώρηση της συνθήκης. Ε, και εφόσον δεν μπορεί να αναθεωρηθεί η συνθήκη, θα πρέπει να λάβουμε τα ρεαλιστικά μέτρα που επιβάλλονται τέλος της παράθεσης. Δηλαδή αν δεν μπορείς να δημιουργήσεις ε, κοινοβούλιο ξεχωριστό για την Ευρωζώνη, τότε εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συσταθεί μια υποεπιτροπή, κάτι τέτοιο. Όπως και κάποιο συνάδελφο από την Κροατία ήταν παρόν και μπορεί να με διαψεύσει αν κάνω λάθο. Είναι σαφέ σε πάση περιπτώσει, ε, τι λέει η γερμανική κυβέρνηση και τι θέση έχει για το μέλλον του ευρώ και της ευρωζώνης. Και θα ήθελα να ρωτήσω, και να το πάω λίγο παραπέρα, διότι εμείς προβληματιζόμαστε ως προς την ενίσχυση της Ευρωζώνης και όλους τους μηχανισμούς που εισάγονται τώρα και θεσπίζονται και στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο και στην Ευρωζώνη. Λοιπόν, αυτό πώς θα επηρεάσει τη μελλοντική πολιτική συνοχής. Έχω μια πολύ απλοϊκή και αφελή ερώτηση και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Θα είναι τελείως διαφορετική η πολιτική συνοχή, ας πούμε, στην Ευρωζώνη σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες εκτός Ευρωζώνης. Τα μέσα και οι μέθοδοι θα είναι διαφορετικά. Και άλλη ερώτηση, συμπληρωματική με την πρώτη. Θυμόμαστε όλοι ότι εδώ και χρόνια έχουμε πρόβλημα με τη λεγόμενη παραδοσιακή πολιτική συνοχή που ήταν συνδεδεμένη με τη σύγκληση και ε, μια πολιτική συνοχή που ευνοούσε τις επενδύσεις, ε, την ανάπτυξη, τη μεγέθυνση οικονομίας, λεγόμενη σύγχρονη πολιτική συνοχή. Ε, ερχόταν σε αντιαδιαστολή με αυτό. Και λέτε ότι ε, δίνεται έμφαση σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Αυτό φαίνεται λίγο σαν οπισθοδρόμηση αν το μελετήσουμε. Γιατί πρόκειται για τη συνοχή, ενώ μακροπρόθεσμα θα γυρίσουμε πίσω και πάλι στη σύγκληση στις μη αναπτυγμένες περιοχές και περιφέρειες και παράλληλα θα έχουμε νέα ε, μέσα για διάφορα επενδυτικά ταμεία που δεν θα είναι εντός της πολιτικής συνοχής, θα είναι κάτι ξεχωριστό. Λάθος το έχω καταλάβει. Είναι πιθανό αυτό το σενάριο. Σήμερα μυρικάζουμε ξανά και ξανά ότι η πολιτική συνοχή είναι η μόνη επενδυτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της ανάπτυξης και της ε, μεγέθυνσης οικονομίας. Όλες αυτές οι αλλαγές θα μας φέρουν πίσω σε μια πολιτική συνοχή ξανά για τους λιγότερο ανεπτυγμένους και τα υπόλοιπα θα πάνε σε άλλο κλάδο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα είναι άλλο για την Ευρωζώνη, άλλο για τις χώρες εκτός Ευρωζώνης. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Γκουτμάνης. Ευχαριστώ, Ντανούτα, για την ευκαιρία που μου δίνεις να μιλήσω. Κύριοι, καλημέρα σας. Σας άκουσα πολύ προσεκτικά, αλλά λυπάμαι πάρα πολύ που θα πω ότι έχω την αίσθηση ότι δεν μπαίνετε σε λεπτομέρειες και χωρίς λεπτομέρειες, χωρίς μαθηματικά και στατιστικές, τα συμπεράσματα που βγάλατε για την Τραπεζική Ένωση, για όλα αυτά τα γενικά που είπατε, δεν είναι αυτό που μας χρειάζεται. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω γιατί επικρίνω τόσο πολύ τέτοιου είδους μελέτες. Um, Έχω στα χέρια μου ε, μια μελέτη της ε, Γενικής Διεύθυνσης ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του κυρίου Βάλτερ Ντέφα με ημερομηνία σημερινή για την ευρωπαϊκή πολιτική κατά την περίοδο 7-13. Και το έχω μελετήσει. Ε, τα γενικά, τα ειδικά, το να κατονομάζεται και να διαπομπεύεται κάποιος κτλ. Και πρέπει να σας πω ότι έχουμε διάφορα στατιστικά στοιχεία Ξέρω την παροιμία που λέει υπάρχουν ε, τα ψέματα, τα χοντρά ψέματα και οι στατιστικές. Αλλά ε, ποια είναι τα πραγματικά αποτελέσματα της ανάλυσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα δικά μου. Και ε, παρόμοια και διαφορετικά, να σας εξηγήσω. Στην ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσπαθούν να φτιάξουν ένα πίνακα που δεν είναι πίνακας διακυβέρνηση χρηστή και ποσοστό απορρόφησης, όπως το γνωρίζετε. Είναι ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο. Και τι βλέπουμε, 7 χώρες από τις 27, είναι μόλις το 25% δηλαδή, έχουν ισχυρή απορρόφηση και καλή διακυβέρνηση. Ασθενή διακυβέρνηση και ασθενή απορρόφηση είναι 9, το 30%, αλλά 20% των χωρών εκατέρωθεν έχουν ισχυρή διακυβέρνηση και ασθενή απορρόφηση ή ασθενή διακυβέρνηση και ισχυρή απορρόφηση. Λοιπόν, ας πάμε στη δική μου ανάλυση να ξεφύγουμε από τις στατιστικές. Προσπάθησα να αναλύσω τα βασικά στοιχεία που συνιστούν την οικονομική διακυβέρνηση. Όταν έχετε υπερβολικό έλλειμμα του προπολογισμού και μακροοικονομικές ανισορροπίες, τα ίδια ισχύουν. Τα γράφει και ο νόμος τώρα και άρχισα να μελετώ από τα ελλείμματα του 9 την απορρόφηση, τις δυνατότητες και το γενικό χρέος. Και τι διαπίστωσα. Δεν θίγω Ρουμανία, Βουλγαρία, που δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν μπόρεσαν να ε, φτάσουν στα συνήθη ποσοστά απορρόφησης. Δεν ξέρω, κανείς δεν μπόρεσε να μου το εξηγήσει, ούτε εδώ στην Κομισιόν, ούτε εθνικές μελέτες, ούτε στα Υπουργεία, ούτε κανείς. Εν πάση περιπτώσει. Ας πάρουμε άλλες χώρες. Παράδειγμα, Ιταλία και Τσεχική Δημοκρατία. Καμία σχέση. Αν δείτε Ιταλία, στο έλλειμμα της θα πηγαίνει πολύ καλύτερα από κάποιες χώρες που έχουν πολύ καλή απορρόφηση. Και από απορρόφηση θα πάει χάλια. Η Ιταλία το 2013 ήταν στην προτελευταία θέση, 26η από 27. Το έλλειμμα του προπολογισμού είναι κάτω του 3%. Εντάξει και το γενικό χρέος τους ε, δεν είναι πολύ ψηλό, αλλά ας το αναλύσουμε. Έχετε τη δυνατότητα να το λύσετε. Ποια είναι τα βασικά επιχειρήματα. Ε, το έλλειμμα του προπολογισμού όχι. Διότι για παράδειγμα υπάρχουν χώρες που έχουν πάρα πολύ χαμηλά ελλείμματα αλλά και κακή απορρόφηση ταυτόχρονα. Βλέπετε τσεχική δημοκρατία. Εντάξει, 3% λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω και είναι το έλλειμμά του. Κριτήρια Μάστριχτ. Αλλά η απορρόφηση είναι χάλια κι αυτή. Είναι να το πάρουμε αντίστροφα. Όχι Εστονία, Λιθουανία που είναι η καλύτερη στην απορρόφηση, αλλά πάμε Ισπανία, Πορτογαλία. Που έχουν και κρίση και ό,τι άλλο θέλετε. Αλλά δεν υπάρχει καμία σχέση. Πώς το συσχετίζεται αυτό. Παράδειγμα, στην Ισπανία το δημόσιο γενικό χρέος είναι 53% το ΕΠ το 9 και 84% το 2012. Τα επίσημα στοιχεία είναι αυτά. Η απορρόφηση όμως δεν είναι κακή. Είναι πέμπτη στην απορρόφηση από 27 χώρες. Και το έλλειμμα του φτάνει 9-10% μέχρι και 11%. Κοιτάξτε τώρα την Πορτογαλία. Τα ίδια. Και ερχόμεθα στο εξή ερώτημα. Και θα πρέπει να γίνει αυτή η ανάλυση. Αλλιώς όλα αυτά τα επιπόλαια, τα επιφανειακά που μας λέτε τι να τα κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Για αυτού που προσπαθούν να πάρουν πολιτικές αποφάσεις. Και να σα εξηγήσω και κάτι άλλο, γιατί τελειώνω με αυτό. Αν δείτε την ανάλυση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα διαπιστώσετε ότι είναι πολύ ενδιαφέροντες οι πίνακοι στην αρχή και πόσο σημαντικά είναι ε, τα χρήματα της συνοχής για διάφορες χώρες. Πήραν τη συνοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Εθνική Χρηματοδότηση Και αν το δούμε σε σχέση με το έλλειμμα, ε, το πραγματικό, διαπιστώνουμε ότι για την Ουγγαρία οι δημόσιες επενδύσεις είναι μέχρι και 95%. Δηλαδή ο μόνος που επενδύει είναι το δημόσιο. Άρα καμία συμπληρωματικότητα. Ξέρετε τι είναι το κρύο αυτό της προσθετικότητας. Ε, το θίξατε. Αλλά για να καταλάβουμε τι γίνεται θα πρέπει να καταλάβουμε ε, τι γίνεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τους υποχρεώνει και στην Λιθουανία 75% πολύ ψηλό. Στην Ισπανία όμως τι γίνεται, 11%. Ή ας πούμε Πορτογαλία πενταπλάσιο, 50%. Τι εννοώ, τι θέλω να πω τελικά. Δεν ξέρω, πάντως τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι δεν είναι εύκολο να βρει κανείς το πραγματικό κλειδί για να ανοίξει αυτή την πόρτα. Για να συνδέσει την πολιτική συνοχή με την απορρόφηση. Και ποσοτικά. Υπάρχει γενική διακυβέρνηση και πώς μπορεί να συνδεθεί. Οι στατιστικές έχουν μεγάλη διασπορά, τεράστια, από 30% και πάνω μέχρι 25% μείον 25%. Ενδεχομένως θα πρέπει να μπει σε μεγαλύτερο βάθος η ανάλυση. Να μην λέμε ότι φταίει το γενικό χρέος, το έλλειμμα, το αρνητικό ισοζύγιο πληρωμών κτλ. Θα πρέπει μαζί να βρούμε, όχι εσείς, μαζί αυτοί που θα κάνουν την επόμενη μελέτη τύπη. Και τελειώνει αυτή η ανάλυση, η, μαθηματική ε, του δίκτυου απορρόφησης, γιατί μαθηματικά μπορεί να έχει πολύ ψηλή απορρόφηση, αλλά αν δείτε την περίοδο, την προηγούμενη την προγραμματική 2000, 2006 ε, και ακόμα πιο παλιά, υπάρχουν χώρες με πάρα πολύ καλή απορρόφηση, που ήταν οι πρώτες που μπήκαν στην κρίση και οι πρώτες που μπήκαν στο δούνο του και ζήτησαν περισσότερα λεφτά. Τεράστια ποσά πήρανε από τη συνοχή. Και αυτό ρωτάω και τους φίλους της συνοχής. Τι τα θέλετε τα λεφτά για τη συνοχή, αφού όταν ξεσπάει η κρίση είστε οι πρώτοι που θα απλώσετε το χέρι ε, και θα ζητάτε λεφτά. Τώρα έχει έρθει η ώρα να πάμε σε πολύ μεγαλύτερο βάθος αγαπητοί κύριοι, διότι αλλιώς τέτοιες αναλύσεις δεν βοηθούν καθόλου στο κοινοβούλιο. Ούτε το σημερινό ούτε το επόμενο. Και θα πρέπει να συνεργαστούμε πολύ περισσότερο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάννης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω τα Σουηδικά εφόσον έχουμε δερμηνία. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο και σας ευχαριστώ πολύ και για τη μελέτη αυτή που μας παρουσιάσατε. Νομίζω ότι θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν χρειαστεί να καθορίσουμε κάποια πράγματα όσον αφορά την πολιτική συνοχή. Είναι πάντως πολύ χρήσιμη η μελέτη αυτή. Εγώ γνωρίζω την εφαρμογή της πολιτικής αυτής στη Σουηδία. Κάπου στη μελέτη λέγεται ότι τα κράτη-μέλη απομακρύνονται όλο και περισσότερο από τη στρατηγική Ευρώπη 2020, ότι κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης χρησιμοποίησαν ουσιαστικά την οικονομική κρίση για να απομακρυνθούν, να πάρουν τις αποστάσεις τους από τη μακροπρόθεσμη αυτή στρατηγική Ευρώπη 2020. Και βλέπουμε ότι οι τοπικοί, οι περιφερειακοί, οι εθνικοί παράγοντες όλο και περισσότερο αναφέρονται σε αυτούς τους μακροπρόθεσμους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Πολύ περισσότερο τελικά τους ακούμε σε περιφερειακό επίπεδο από ό,τι σε εθνικό επίπεδο, από ό,τι στα κράτη-μέλη. Κάθε φορά που διαπραγματευόμαστε όμως συμφωνίες, φαίνεται ότι τα κράτη-μέλη και οι κυβερνήσεις τους αποφασίσουν τελικά να απομακρυνθούν από τη στρατηγική αυτή, χρησιμοποιώντας ως βασικό επιχείρημα για να κάνουν κάτι τέτοιο τις νέες συνθήκες που έχουν προκύψει από την οικονομική κρίση, το γεγονός ότι δεν μπορούν να διχειριστούν όπως το παρελθόν τα δημόσια οικονομικά. Τι μπορείτε να μας πείτε εσείς προς αυτό, τουλάχιστον έτσι βλέπω εγώ τα πράγματα στη Σουηδία. ότι ε, υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη που διατρέχουν σαστικά αυτόν τον κίνδυνο. Δεν ξέρω αν άλλα κράτη-μέλη λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας απαντήσετε σε σχέση με αυτά. Ευχαριστούμε κυρία Μαλέτιτς. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω ότι η ανάλυση αυτή καταδεικνύει ξεκάθαρα ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών. Το πρόβλημα είναι ότι χρειάζεται μεγαλύτερο συντονισμό των διαφόρων πολιτικών. Και το βλέπω το πρόβλημα αυτό και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, ΕΚΟΝ, και στην Επιτροπή αυτή συζητάμε συνεχώς διάφορα μέτρα που έχουν να κάνουν με το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Εξάμεινο. Συζητάμε όλο και περισσότερο τη διαδικασία δημοσίου ελλείμματος, τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, τις ειδικέ αναχώρασεις τάσει και προσπαθούμε να προωθήσουμε ευνοϊκά προγράμματα εθνικών μεταρρυθμίσεων τα οποία θα πρέπει να έχουν ως στόχο την μείωση του δημοσίου ελλείμματος και την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης. Καταλαβαίνετε ότι τα ζητήματα αυτά έχουν άμεση σχέση με την πολιτική συνοχή και παρόλα αυτά συζητώνται εντελώ ξεχωριστά από την πολιτική συνοχή. Τα εθνικά λοιπόν αυτά προγράμματα, καθώς επίσης και η πολιτική συνοχή θα πρέπει να αντικατοπτρίζει πλέον τις ειδικές αναχώρα συστάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά βλέπουμε ότι μόνο η Γενική Διεύθυνση Προπολογισμών, το ΕΚΟΦΗΝΑ η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή κάποιοι υπουργοί μεμονωμένα τελικά συζητούν τα ζητήματα αυτά. Και από την άλλη έχουμε άλλες επιτροπές όπως τη δική μας, την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, η οποία συνεργάζεται με υπουργού αρμόδιους για την περιφερειακή ανάπτυξη σε διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις λαμβάνουν καλύτερες, περιπτώσεις, ε, καλύτερες αποφάσεις, με σε ορισμένα κράτη-μέλη από ό,τι σε άλλα και παράλληλα με όλα αυτά έχουμε και συγκεκριμένα προγράμματα και στρατηγικά έγγραφα για την πολιτική συνοχής και ουσιαστικά δεν βλέπω να υπάρχει μία διασύνδεση, μία ισχυρή σχέση ανάμεσα σε όλες αυτές τις διαφορετικές πολιτικές, τις διαφορετικές συμφωνίες και πολιτικές που προωθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και που άμεσα τελικά συνδέονται με την πολιτική συνοχής και παρόλα αυτά συζητώνται εντελώ ξεχωριστά. Αναφέρομαι σε διαδικασίες ε, όπως ε, η αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, αναφέρομαι στις ειδικέ αναχώρα συστάσεις, αναφέρομαι σε διαδικασίες ε, οικονομικές που εφαρμόζονται σε κράτη-μέλη που προσπαθούν να καταπολεμήσουν το περιβολικό έλλειμμα και ουσιαστικά καθότι ε, παράλληλα διεξάγονται όλες αυτές οι συζητήσεις, κάποια κράτη-μέλη δεν μπορούν να καταλάβουν τελικά αν υπάρχει μια γενική ενωσιακή προσέγγιση. Αυτό το βλέπω για παράδειγμα έντονα στην Κροατία, η οποία πρόσφατα προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία καλείται αυτή τη στιγμή να λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις και να εφαρμόσει συγκεκριμένες πολιτικές. Για παράδειγμα, αν μειωθούν οι μισθοί στην Κροατία, επηρεάζεται και η ανταγωνιστικότητα της χώρας, αν μειωθούν μισθοί και συντάξεις, αυξάνονται τα ποσοστά ένδια στη χώρα, επομένως επηρεάζονται και οι απότεροι στόχοι της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020. Ουσιαστικά οι μισθοί και οι συντάξει είναι το μεγαλύτερο τμήμα των δημοσίων δαπανών μα. Και βλέπουμε ότι περισσότερε αποφάσει που λαμβάνονται έχουν να κάνουν τελικά με κεφαλαιακέ επενδύσει και ουσιαστικά βλέπουμε ότι οι επενδύσεις αυτές όλο και περισσότερο μειώνονται και αυτό με τη σειρά του επηρεάζει την ε, δυνατότητά μας να χρησιμοποιήσουμε την πολιτική συνοχή. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να βρεθούν κάποιες λύσεις για να καταφέρουμε να υποστηρίξουμε τις χώρες εκείνες οι οποίες έχουν ε, ένα επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης κατώτερο του 75% σε σχέση με τον ευρωπαϊκό όρο, γιατί ξέρετε ότι η πολιτική συνοχή τελικά στις χώρες αυτές επικεντρώνεται και θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στις χώρες αυτές να ανασάνουν, για να το πω έτσι. Δηλαδή, αν βρίσκονται στη δικασία υπερβολικού ελλείμματος, να μπορούν αν μη τι άλλο να έχουν ένα περιθώριο ευελιξίες για να κάνουν επενδύσεις. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέμε ότι οι χώρες αυτές μπορούν να υπερβούν τελικά το 3% όσον αφορά το δημόσιο έλλειμμά τους, αν οι επενδύσεις αυτές οι δημόσιες προωθούνται έχουν τη μορφή συγχρηματοδότησης προγραμμάτων πολιτικής συνοχής, γιατί οι επενδύσεις αυτές ουσιαστικά έχουν ως στόχο να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη. Αν μειωθεί, αν απαιτούμε εμεί τη μείωση της συγχρηματοδότησης, καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο που οδηγεί σε μειωμένη οικονομική ανάπτυξη τελικά. Πρόεδρος, θα ήθελα να πάρει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Κατερίνα Ρουμπιάνης είναι μαζί μας. Έχετε το λόγο. Θέλετε μάλλον να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τους συντάκτες της έκθεσης για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Πραγματικά μας δίνει πολλές αφορμές για να προβληματιστούμε και να θέσουμε νέα ερωτήματα. Για το πώς θα διαμορφωθεί μια νέα πολιτική συνοχής με την αργά εξελισσόμενη οικονομική διακυβέρνηση. Υπάρχουν θέματα τα οποία καλό ήταν να τα σκεφτούμε περαιτέρω και προσεκτικά. Απλώς θέλω να σταθώ σε τρία σημεία. Πρώτον, όταν η μελέτη αναφέρεται στο ότι υπάρχει ε, μεγάλος κίνδυνος υψηλότερης, σε χώρες με μεγάλα ποσοστά χρέους, να υπογραμμίσω εδώ ότι τουλάχιστον ως τώρα δεν βλέπουμε να υπάρχει σαφή συσχετισμό μεταξύ των δύο. Υπάρχουν χώρες που έχουν πιεστεί σοβαρά από τα προγράμματα προσαρμογής όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία αλλά έχουν από τους καλύτερους δείκτες ε, απορρόφησης στην ε, τελευταία περίοδο προγραμματισμού. Αυτό μας κάνει να φανταστούμε ότι οι σημαντικές δημοσιονομικές πίεσεις δεν ε, συνιστούν απαραίτητα παράγοντα χαμηλότερης απορροφικότητας. Έπειτα, ο συσχετισμός μεταξύ του υψηλού επίπεδου χρέους και της επιβολής κυρώσεων βάσει των ε, νέων κανόνων για τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα. λόγω του δημοσιονομικού ελλείμματος ή του υψηλού χρέους δεν ε, ενεργοποιούνται απαραίτητος αυτόματα κυρώσεις όταν δεν υπάρχει πραγματική δράση μετά από συστάσει του Συμβουλίου, τότε επιβάλλονται ε, κυρώσει και τότε ενεργοποιείται ο μηχανισμό. Σε κάθε περίπτωση όμω η του υψηλου χρεους δεν ενεργοποιουνται απαραιτητος αυτοματα κυρωσεις οταν δεν υπαρχει πραγματικη δραση μετα απο συστασεις του συμβουλιου τοτε επιβαλλονται ε κυρωσει και τοτε ενεργοποιειται ο μηχανισμος σε καθε περιπτωση ομως η αρση της χρηματοδότησης έχει να κάνει και με συγκεκριμένα όρια και με πρόσθετες συστάσεις. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο, ξέρετε, ότι ούτω ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προηγουμένω θα δημοσιεύσει κατευθυντήριε γραμμέ για να εξηγήσει πώ η μακροοικονομική αιρεσιμότητα θα εφαρμόζεται ακριβώ. Και τρίτον, και τελευταίο για την ώρα, είναι ότι η μελέτη αναφέρει ότι υπάρχει ενδεχόμενο κίνδυνο επικέντρωση σε συγκεκριμένου τομεί τη πολιτική όπω θα τη χαράξουμε. Σε αυτή τη φάση, ο συσχετισμό που υπάρχει βάσει του άρθρου 5 διατηρεί την αρχή των εταιρικών σχέσεων ω μια από τι κυρίαρχε αρχέ τη πολιτική συνοχή. Είναι τουλάχιστον τόσο ισχυρή όσο και στο παρελθόν. Οπότε, όταν διαπραγματευόμαστε εταιρικέ ε, συμφωνίε, προγράμματα συνεργασία με οικονομικού φορεί, με φορεί των ε, πόλεων, των αστικών κέντρων, των περιφερειών και επαρχιών, Πρέπει να είναι πολύ σαφής ε, η όρη εκτέλεση των λειτουργικών αυτών προγραμμάτων. Πρόεδρος, δεν ζητά άλλο κανεί το λόγο. Να εκμεταλλευτώ και εγώ αυτή την ευκαιρία για να πω λίγα λόγια. Να θυμίσω σε όλους μας την ιστορία αυτές τις μελέτες Αλλά πρώτα ο Γιώχημ Τσέλερ, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ζήτησα το λόγο μόνο γιατί άκουσα το Γιάνν Όλμπριχτ που ερμήνευσε έτσι τα λόγια του κυρίου Σόιπλε ότι θέλει η γερμανική κυβέρνηση ένα ξεχωριστό κοινοβούλιο για την Ευρωζώνη. Ε, θέλω να το διαψεύσω αυτό. Κανείς στη Γερμανία δεν επιθυμεί ξεχωριστό κοινοβούλιο για την Ευρωζώνη. Μην ανησυχείτε. Αυτό που θέλουμε εμείς όμως είναι να υπάρχει μια συμφωνία, μια συνεννόηση μεταξύ των κρατών που είτε είναι εντός της Ευρωζώνης είτε ε, προσδοκούν την ένταξή τους και σε εθνικό επίπεδο να συντονίζονται με τα όσα συζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λέει επίσης ο Γερμανός Υπουργό Οικονομικών ότι εκείνα τα κράτη που δεν είναι πρόθυμα ε, να μπουν στο ευρώ, μακροπρόθεσμα, δηλαδή το έχουν αποκλείσει για τους αυτούς τους, ε, τότε δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση. Περί αυτού πρόκειται. Οι χώρες όμως που είναι μέλη τη Ευρωζώνη και εκείνε που μέσω ή μακροπρόθεσμα φιλοδοξούν να ενταχθούν, χρειάζονται κάποιες δομέ για να συντονίζονται οι εθνικές αποφάσεις που λαμβάνονται στα εθνικά κοινοβούλια σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για χώρε μέλη τη Ευρωζώνη σημερινά ή μελλοντικά. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να είναι ε, επιτροπή τη Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Αυτό είναι ακόμα προ συζήτηση. Μεταξύ μα θα το συζητήσουμε. Απλώ για να σα καθησυχάσω. Κανεί δεν επιθυμεί ξεχωριστό κοινοβούλιο για τι χώρε τη Ευρωζώνη. Εάν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, λοιπόν, να πω και εγώ δύο λόγια. Τα εξή. Πέρσι τον Ιούνιο, πρότεινα να χρησιμοποιήσουμε το τελευταίο περιθώριο που είχαμε, το τελευταίο μερίδιο για έκθεση ίδιας πρωτοβουλία για τη σύνταξη μιας έκθεσης ίδιας πρωτοβουλίας ακριβώς από το θέμα αυτό το συσχετισμό μεταξύ των αλλαγών στη μακροοικονομική διακυβέρνηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον τη πολιτική συνοχή. Υποτίθεται ότι θα δημοσιευόταν και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περίπου τον Νοέμβριο μια ανακοίνωση για το θέμα αυτό, αλλά αυτή ε, ξανεμίστηκε, ξαϊλώθηκε τελείω από το πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2013. Οι συντονιστέ και η Επιτροπή εν τη Σοφία του αποφάσισαν να μην ε, συνταχθεί τέτοια έκθεση ιδία πρωτοβουλία και να αφιερώσουμε αυτό το μερίδιο σε μια άλλη ε, πρωτοβουλία. Τουλάχιστον όμως έχουμε αυτή τη μελέτη για να το αφήσουμε αυτό σκληροδότημα για τη Μελλοντική Επιτροπή Περιφερειών. Διότι το 2013 και 2014 με τις αλλαγές στην οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που προέκυψε από τη σκοπιά της πολιτικής συνοχής φαίνεται να υπάρχουν σοβαροί συσχετισμοί μεταξύ της συνοχής και της οικονομικής ακριβώς διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως διαμορφώνεται. Οπότε πραγματικά χρειαζόμασταν ένα τέτοιο ε, κληροδότημα, μια τέτοια κληρονομιά για την ερχόμενη Επιτροπή. Το ε, μελλοντικό Ευρωκοινοβούλιο στην αξιολόγηση της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να αλλάξει δραστικά την ε, οπτική του γωνία. Δεν θα κοιτάζει μόνο τι κάνουν τα μέλη τα κράτη-μέλη, οι περιφέρειες και τα αστικά κέντρα στην αξιολόγηση, στην αποτίμηση, το να δει τα ποσοστά απορρόφησης, τις προσπάθειές τους. Δεν θα αρκεί να βλέπει μόνο την πολιτική αυτή απομονωμένα, αλλά όπως φαίνεται και από την έκθεση και τις ε, συστάσεις της, το Ευρωκοινοβούλιο και ιδίως αυτή η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζουν την πολιτική συνοχής εντός του ε, πλαισίου του τοπίου της ε, εκπόνησης της μέσα σε ένα ευρύτερο ε, τοπίο οικονομικής δικυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντί λοιπόν να κοιτάζουμε μόνον κράτη-μέλη ή περιφέρειες, θα πρέπει στο Ευρωκοινοβούλιο να εξετάζουμε προσεκτικά μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το πώ καταρτίζουν την ε, οικονομική του διακυβέρνηση, την οικονομική διακυβέρνηση γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν δούμε και το οικονομικό κόστο, όπω προκύπτει από τη χρηματοπιστωτική και οικονομική ένωση, με συγκεκριμένη μυθοδολογία που προκύπτει, ή την πρακτική τη επιβολή κυρώσεων εντό των όσων έχουν ονομαστεί προσωρινά μακροοικονομική ρεσιμότητα, θα πρέπει λοιπόν να έχουμε και αυτά κατά νου όταν εξετάζουμε την πολιτική συνοχή. Να δούμε τι κάνουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ώστε να μην υποβαθμιστεί αυτή η πολιτική σε ένα απλό εργαλείο ε, υλοποίηση τη οικονομική διακυβέρνηση και άλλων παραλληλών στόχων. Ούτε και να τιμωρηθούν άδικα κάποιοι για σφάλματα που προκύπτουν από άλλες πολιτικές. Βρίσκω λοιπόν ότι αυτό το συμπέρασμα είναι άκρος ε, σημαντικό για μας. Να σκεφτούμε πώς πρέπει να αλλάξουμε και εμείς την αντιμετώπιση μας, τον ρόλο της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής και πώς μπορούμε να διοργανωθούμε καλύτερα στη συνεργασία μας εντός του Ευρωκοινοβουλίου. Η συνεργασία με τις Επιτροπές Οικονομικών Υποθέσεων, ή προπολογισμών είναι ζωτική σημασία. Θα πάρει διαφορετική μορφή από αυτή που σήμερα γνωρίζουμε. Αυτό που προκύπτει λοιπόν από την έκθεση δεν είναι πάρα πολύ αισιόδοξο για το Ευρωκοινοβούλιο, διότι αφήνεται την υπόνοια ότι μπορεί και να παραγωνιστούμε από την όλη διαδικασία όπως θα διαμορφωθεί στο μέλλον. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν σοβαρά πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις στο μέλλον, διότι από το 2014 έως το 2020 ξεκινά μια νέα εποχή πραγματικά για την πολιτική συνοχή. Και από τη μια είμαστε υπερήφανοι, διότι καταφέραμε ως τώρα να ε, φτιάξουμε πραγματικά την καταξοχήν επενδυτική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Την συμπεριλάβαμε στην οικονομική διακυβέρνηση στο πρώτο μέρο τη μακροοικονομική αρισιμότητα, αλλά υπάρχει και ένα κόστος, ένα τίμημα που πρέπει να καταβάλουμε και κάποιοι κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπιστούν από τώρα. Να πω λοιπόν ότι ο στόχο δεν ήταν να δούμε την διακυβέρνηση τη πολιτική στην παραδοσιακή της έννοια, πώ ασχολούμαστε με τα θέματα χειρισμού τη πολιτική κατά την υλοποίησή τη, αλλά να δούμε την πολιτική αυτή Εντό ενός μεταβαλλόμενου μοντέλου οικονομική διακυβέρνηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή ήταν η δική μου συμβολή στη συζήτηση. Εάν θέλετε να σχολιάσετε κι εσείς παρακαλώ. Ή Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να δώσω μια απάντηση που θα μπορούσε να απαντά ταυτόχρονα σε πολλές από τις παρατηρήσεις που έγιναν για το θέμα της διαφοροποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αλλαγής της κατά πρώτο. Νομίζω ο κ. Σόλμπριχτ και αυτό μίλησε. Η πολιτική συνοχής, αναμφισβήτητα, είναι πολιτική της Ευρώπης των 28. Έτσι έχει συμπεριληφθεί αυτό και στη συνθήκη. Έτσι έχει καταγραφεί. Αυτό όμως που αρχίζουμε να βλέπουμε είναι ότι καθώς η Ευρωζώνη ε, των 18 συν οι άλλοι δύο που θέλουν να, να πάρουν μέρος ε, σε πρωτοβουλίες οικονομικής ένωσης, καθώς αυτοί συγκλίνουν περισσότερο, βλέπουμε κάποιες πολιτικές με στόχους συνοχής να επηρεάζονται από διάβλους που δεν έχουν να κάνουν με τη συνοχή. Αυτό προσπαθούσα να πω. Γι' αυτό και ε, το κατά πόσο αυτά που λέτε με τον κύριο Τσέλερη όχι ισχύουν μπορούμε να το δούμε αργότερα. Αλλά ασχέτως με το αν υπάρχει νέα θεσμική οργάνωση, επιτροπή ή ένα ε, νέο κοινοβούλιο για την Ευρωζώνη, υπάρχουν πολιτικές οι οποίες θα αφορούν μόνο ένα υποσύνολο των κρατών μελών. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα νομιμοποίησης και ελέγχου παρακολούθηση για του κυβερνητικού φορεί που θα τα παρακολουθούν αυτά. Αυτό είναι και το ζουμί όσων προσπαθούσαμε να πούμε με όλα αυτά τα ε, σχόλια και τι ε, σκέψεις που αναπτύξαμε. Στενότερο συντονισμό θα υπάρχει, αλλά κάποιε φορέ θα υπάρχει συντονισμός εντός, εκτός και επί τα αυτά. Δεν θέλω να υπερασπιστώ τη χώρα από την οποία προέρχομαι, αλλά ναι, νομίζω είστε την Κροατία. Υπάρχει κατά δεύτερον και μια δυσκολία την οποία προκαλούν ακριβώς οι αλλαγές στην οικονομική διακυβέρνηση. Το πώς θα συμφιλιώσουμε τους στόχους της μακροοικονομικής πολιτικής με τη συνοχή. Τα είπατε πολύ καλά. Βρήκατε το σχετισμό. Διότι υπάρχει ένταση μεταξύ των στόχων της Ευρώπης το 2020 και των στόχων μακροοικονομικής σταθερότητας. Αλλά πέραν αυτού τα εθνικά κοινοβούλια που μπορεί να βλέπουν τον εαυτό τους ως ε, κυρίαρχα σε θέματα δημόσιου προπολογισμού. Εκεί μπορεί να χάνουν αυτήν τους την ε, αναμφισβήτητη ως τώρα αρμοδιότητα. Εκεί έχουμε θέμα λογοδοσίας και νομιμοποίησης στην περίπτωση των προτάσεων για την πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση. Τώρα το πώς θα χειριστούμε αυτή την ένταση, πώς το Ευρωκοινοβούλιο εντάσσεται σε αυτό το τοπίο έντασης, είναι κάτι πολύ αβέβαιο ακόμη. Νομίζω το Κοινοβούλιο θα πρέπει να προτείνει εκείνο πρωτοβουλίε για να αντιμετωπίσει αυτού τα προβλήματα, τα οποία δεν νομίζω ότι ακόμη τα γνωρίζουμε αρκετά. Η κυρία Χούμπνερ ε, έχει δίκιο. ε, Όντω έγινε μια νέα χάραξη τη πολιτική συνοχή ω τη καταξοχήν επενδυτική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά υπάρχουν και πολύ σοβαροί περιορισμοί. Δεν μπορούμε να κοιτάζουμε τα ποσοστά απορρόφηση του 2009 για να δούμε τι θα γίνει το 2013 και μετά. Ε, ένα τελείω νέο σενάριο αναπτύσσεται πλέον καθώ η πολιτική συνοχή αλλάζει. Βεβαίω τα ποσοστά απορρόφηση δεν μπορούν ε, αμέσω να συσχετίζονται με το τι συμβαίνει στα δημοσιονομικά ενός κράτους. Υπάρχει και η δημόσια δίκηση, υπάρχει η άσκηση ελέγχου. Κάποια από αυτά έχουν να κάνουν με τις διαφορές μεταξύ του επίπεδου της Επιτροπής, των εθνικών κρατών, των περιφερειών, των, της έντασης των ελέγχων, του κατά πόσο οι κανόνες ακολουθούνται εφαρμόζονται νόμοι και το καθεξής. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι μπορούμε να αξιολογήσουμε την ε, παρελθούσα ε, πολιτική συνοχής για να βγάλουμε συμπεράσματα για το μέλλον. Προσπαθούμε να φανταστούμε ότι θα γίνει αναδρομική, πάντως αξιολόγηση της πολιτικής συνοχής δεν θέλαμε να κάνουμε με αυτή την έκθεση. Και να δώσω τώρα το λόγο και στον Τζον για να σχολιάσω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you. Ε, Ευχαριστώ. Να προσθέσω κι εγώ κάποια σημεία σε αυτά που είπε ο Ιαν όσον αφορά τα σχόλια του Γιάννου Όλμπριχτ για τη μελλοντική σχέση ανάμεσα στα νέα μέσα και τη μορφή που θα πάρει πολιτική συνοχή σε σύγχρονη παραδοσιακή. Κοιτάξτε, εξαρτάται από την μελλοντική μορφή που θα έχουν άλλα αντιτιθέμενα στην πολιτική συνοχή μέσα αν θα καλύπτουν δηλαδή όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση όχι, αν θα υπάρχουν ε, θεματικές προτεραιότητες. Πάντως ενδεχομένως να έχουμε τελικά ένα νέο μέσο το οποίο θα έχει ως στόχο να προωθεί περισσότερο μία εδαφική εξισορρόπηση και η οποία θα βασίζεται περισσότερο σε συγκεκριμένε επενδύσεις που θα μπορούν να γίνουν σε συγκεκριμένε περιφέρειες και οι οποίες θα συνδέονται με διάφορους στόχους όπως η αντιμετώπιση του ελλείμματος, η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της καινοτομίας και το καθεξής. Μπορούμε να δούμε το παράδειγμα το γερμανικό που δεν είναι το καλύτερο για το ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά σε περιφερειακό επίπεδο όντως λειτουργεί πάρα πολύ αποτελεσματικά και τελικά εξισώνει κάπως τις περιφέρειες μεταξύ τους με τη θετική έννοια. Υποστηρίχθηκαν για παράδειγμα κάποιες περιφέρειες της Ανατολικής Γερμανίας που υστερούσαν σε σχέση με τη Δυτική Γερμανία ή γίνουν επενδύσεις σε συγκεκριμένα λάντερ, κρατήδια. Όσον αφορά τώρα τα ερωτήματα του κυρίου Γκοτμάνης, Συμφωνώ με το θεμελιώδες αυτό ερώτημα το οποίο τίθεται. Πώς διαφοροποιούνται τα διάφορα ποσοστά απορροφήσεις από τη μία περιφέρεια στην άλλη. Ακόμα δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς. Έχουν γίνει διάφορες μελέτες οι οποίες λένε ότι είναι τελικά οι περιφερειακές διοικητικές ικανότητες αυτές οι οποίες καθορίζουν το ποσοστό απορρόφησης, αλλά τι είναι τελικά περιφερειακή διοικητική ικανότητα και πώς γίνεται κάποιες ε, χώρες που έχουν ισχυρές κυβερνήσεις σε τοπικό επίπεδο να έχουν χαμηλά επίπεδα απορρόφησης και το αντίστροφο. Έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια στοιχεία, για παράδειγμα χώρες με ανίσχυρη ε, διακυβέρνηση, με αδύναμη διακυβέρνηση, έχουν πολλές φορές κάποιους περιφερειακούς θύλακες που έχουν πολύ καλά επίπεδα διοικητικής ικανότητος σε σχέση με την κεντρική κυβέρνηση. Από την άλλη ξέρουμε ότι υπάρχουν και χώρες με πολύ ισχυρή κεντρική κυβέρνηση που παρόλα αυτά υστερούν σε περιφερειακό επίπεδο. Δεν υπάρχουν δηλαδή σε περιφερειακό επίπεδο οι απαραίτητες διοικητικές δυνατότητες προκειμένου να προωθηθεί εκεί σωστά η πολιτική συνοχής. Δυστυχώ δεν μπορέσαμε στη δική μας την ε, μελέτη να καλύψουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Τώρα, ένα ακόμα ερώτημα το οποίο ακούστηκε ήταν το ότι, ε, μάλλον ο λόγος για τον οποίο απομακρύνονται τα κράτη-μέλη από την στρατηγική Ευρώπη 2020 χρησιμοποιώντας το πρόσχημα τη δικαιολογία της οικονομικής κρίσης. Κοιτάξτε, αυτό βρίσκεται τώρα στο κέντρο των διαπραγματεύσεων που γίνονται μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα οποία προσπαθούν να επικεντρώσουν κάποιες επενδύσεις στα πλαίσια της Ευρώπης 2020 ή ζητάνε μερικές φορές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τους δώσει την απαραίτητη ευελιξία για να έχουν μια πιο σφαιρική προσέγγιση όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταλάβουμε κάπως τις ανησυχίες των κρατών μελών. Μιλούσαμε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Ελλάδας, οι οποίοι μου λέγανε ότι δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να προωθήσω την ιδέα της ευφυούς εξειδίκευσης και τις σχετικές επενδύσεις όταν υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες δεν ξέρουν καν αν θα υφίστανται τους επόμενους έξι μήνες, αν θα έχουν χαροκοπήσει ή όχι. Νομίζω λοιπόν ότι σαφώς κάποιες επιλογές πρέπει να γίνουν και στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα του συντονισμού, για άλλη μια φορά, νομίζω ότι πάλι σε εθνικό επίπεδο, ανακράτος μέλος πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Σε ορισμένα κράτη-μέλη έχουμε το Υπουργείο Οικονομικών που είναι η αρχή τελικά για το συντονισμό της πολιτικής συνοχής και στι χώρε συνήθω αυτέ η πολιτική συνοχή αντιστοιχεί σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των δημοσίων επενδύσεων και υπάρχουν στι χώρε αυτέ πολύ έντονε διασυνδέσει ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών ή άλλου εθνικού φορεί και το ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε άλλε πάλι χώρε βλέπουμε ότι υπάρχουν Υπουργοί Οικονομικών που δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την πολιτική συνοχή και τι σχετικέ επενδύσει. Γιατί ακριβώ οι επενδύσει αυτέ αποτελούν πολύ μικρό ποσοστό των δημοσίων επενδύσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να πλαισιώσουμε όμως σωστά τις διαπραγματεύσεις αυτές και να καταφέρουμε να διασυνδέσουμε τελικά την πολιτική συνοχής με τους στόχους της μακροοικονομικής πολιτικής. Και έπειτα η διαδικασία υποβολή αναφαρών και γενικότερη λογοδοσία. Ποιο θα είναι το σύστημα αυτό το οποίο θα προκύψει προκειμένου να έχουμε μια πιο, ένα πιο αυστηρό πλαίσιο λογοδοσία από τα κράτη-μέλη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των κοινοτικών πόρων στα πλαίσια τη πολιτική συνοχή. Μια τελευταία παρατήρηση όσον αφορά τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προφανώς αποδεχόμαστε ότι η διασύνδεση ανάμεσα στα υψηλά επίπεδα χρέους και τις κυρώσεις για την πολιτική συνοχή έχει να κάνει με το ποσοστό συμμόρφωση σε σχέση με τις διορθωτικές δράσεις και προφανώς εμείς σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε η διασύνδεση αυτή, ο συσχετισμός αυτός να γίνει ακόμα πιο αυστηρός. Ουσιαστικά αυτό το οποίο θέλαμε να πούμε στη μελέτη μας είναι ότι οι χώρες εκείνες οι οποίες θα επηρεαστούν περισσότερο από τα επίπεδα χρέους και από τα σχετικά επίπεδα επενδύσεων στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής είναι κυρίως οι χώρες αυτές οι οποίες βρίσκονται σε συγκεκριμένα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής και έπειτα έχουμε και όλες τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στα πλαίσια του ρυθμιστικού πλαισίου. Ακριβώς επειδή η οικονομική διακυβέρνηση έχει αλλάξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε πάρα πολλές χώρες, έχει μειωθεί και ο ρόλος των εταίρων εκείνων που είχαμε στο παρελθόν, όπως η τοπική αυτοδιοίκηση, οι τοπικοί φορείς. Βλέπουμε ότι η συμμετοχή τους διαφέρει πάρα πολύ από τη μία χώρα στην άλλη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ομάδα που το ε, εκπώνησε, γιατί είμαστε σε αχατογράφητα ύδατα και άγνωστο έδαφος και εξετάσατε την πολιτική συνοχή στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης ε, σίγουρα θα υπάρχουν ακόμα πολλά να γίνουν ε, σε περισσότερες λεπτομέρειες στο μέλλον σε άλλες μελέτες. Σας ευχαριστώ πάντως την ομάδα που εκπονήσατε ε, αυτή τη μελέτη και τους δύο καθηγητές και όλους τους ενεχομένους αυτή την προσέγγιση και την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα Ελπίζουμε να έχει έρθει ο Γενικός Διευθυντής, κύριος Βάλτερ Ντέφα. Εδώ πρέπει να έρθείτε. Άλλο καθηγητές, άλλο υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Yeah. experts around and uh, no, you I'm want anybody. You can. You, you are invited. If you want to sit with, uh, have somebody else, you are, you're welcome. Anybody from the Commission that would like to. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όποιο θέλει να έρθει να καθίσει δίπλα στο Γενικό Διευθυντή, παρακαλώ. Είστε πρόσδεκτοι. And I would like to, to welcome Walter Defa. Καλώς ορίζω τον κύριο Βάλτερ Ντέφα. Εδώ γράφει Γενική Διευθυντή Δέγγιο. Ποιο είναι το νέο ακρονίμιο τώρα, γιατί μπήκε και η αστική διάσταση, έχει αλλάξει η Γενική Διεύθυνση. Ε, ο κύριος Βάλτερ Ντέφο είναι Γενικός Διευθυντής της νέας πλέον Γενικής Διεύθυνσης και συμπεριλαμβάνει και την αστική διάσταση και στον τίτλο. Ε, θελήσαμε να σας καλέσουμε για να μάθουμε πού βρισκόμαστε λίγο Τι έγινε στην περίοδο 2007-2013, είμαστε πιο πολύ στραμμένοι προς το μέλλον, να κάνουμε και έναν απολογισμό λίγο ε, της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ Ντανούτα για την πρόσκληση αυτή να μιλήσω εδώ και να συζητήσουμε μαζί ε, για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής στην προγραμματική περίοδο 7-13, που πλέον θεωρείται παλιά περίοδος <laughs> αφού έληξε. Και όπως είπατε γνωρίζουμε όλοι ότι δεν έχει λέξει καθόλου. Ε, τώρα, τι θέλω εγώ να κάνω, να σας πω. Να σας ενημερώσω για τα αποτελέσματα και ε, τι έχει προκύψει από την πολιτική, όπως αυτή εφαρμόζεται. Έχετε τη στρατηγική έκθεση που παρουσιάζεται τον Απρίλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο μεταξύ έχουμε μερικά νέα στοιχεία και δεδομένα. Η στρατηγική έκθεση βασίστηκε μέχρι το 2011 στα στοιχεία και τώρα πλέον έχουμε και στοιχεία μέχρι τα τέλη του 2012. Και στη συνέχεια θα μπω σε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς η πολιτική ανταποκρίθηκε και απάντησε στην κρίση. Γιατί κυριάρχησε αυτό το γεγονός στη συγκεκριμένη περίοδο. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση χτυπήθηκε από τη χειρότερη κρίση που έχει γνωρίσει ποτέ από τη σύστασή της. Και Κάτι άλλο που θα σας ενδιαφέρει όλους στην Επιτροπή σας είναι πού βρισκόμαστε από πλευράς απορροφητικότητας. Θα σας δώσω τα τελευταία στοιχεία που έχουμε. Το θέμα που μας ενδιαφέρει όμως και είναι κρίσιμο στην πολιτική μας δεν είναι μόνο η απορροφητικότητα αλλά και η οικονομική διαχείριση που είναι αλληλένδετα αυτά μεταξύ τους και θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι δαπάνες που κάνουμε είναι νόμιμες και ε, σωστές. Και ένα τελευταίο που έχει επίση πολύ μεγάλη σημασία, θέλω να σας ενημερώσω για τις υποστηρικτικές δράσεις που αναλαμβάνουμε τώρα ε, σε μεγαλύτερη ένταση από ό,τι στο παρελθόν για να υποστηρίξουμε τη διοικητική ικανότητα ε, και τις δυνατότητες των περιφερειών και των κρατών μελών που αγωνίζονται και παλεύουν για να εφαρμόσουν την, την πολιτική αυτή και να τη διαχειριστούν οικονομικά. Λοιπόν, η πολιτική συνοχής αποδίδει, έχει αποτελέσματα και εν μέσω κρίσης. Όταν κάναμε τα μοντέλα μας, τι κάναμε. Και αυτό έχει να κάνει και με την κρίση. Για τους βασικούς δικαιούχους, κατά τη διάρκεια των ετών, η πολιτική τους έχει επηρεάσει τουλάχιστον κατά ε, μία ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ. Έχει αυξηθεί. Μπορεί να φαίνεται λίγο αυτό, αλλά και το ΑΕΠ είναι μεγάλο μέγεθος και το 1% του ΑΕΠ επίσης μεγάλο είναι και ε, χρειάζονται και μεγάλες προσπάθειες. Ε, μέχρι εκεί. Αν δεν υπήρχε η κρίση θα ήταν πιο μεγάλη αποτελεσματικότητα προφανώς των ταμείων. Ο ρυθμός μείωσης των διαφορών ε, κατά τη διάρκεια των ετών με την κρίση σταμάτησε και αντιστράφηκε. Δηλαδή με την κρίση αυξήθηκαν οι ε, διαφορές. Και αυτό ανησυχεί τους ενδιαφερόμενους και εκείνους που ασχολούνται με την περιφερειακή πολιτική. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, βάλαμε κάποια βασικά επιτεύγματα της περίοδου. Είναι μέχρι το τέλος του 2012, όπως σας είπα. Είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν για επιχειρήσεις, startup, ε, νεότευκτες και νεοσύστατες που ε, υποστηρίζονται αυτοκινητόδρομοι, σιδηρόδρομοι, ε, ε, ε, φτιάχτηκαν 5 εκατομμύρια πολίτες έχουν πρόσβαση σε ευρωζωνικό διαδίκτυο, 3,2 εκατομμύρια έχουν επιπλέον πρόσβαση σε πόσιμο νερό καθαρό, στο κοινωνικό ταμείο έχουμε 15 εκατομμύρια συμμετέχοντες στο χρόνο και στα χρηματοδοτικά μέσα έχουμε 940 τέτοια και είναι σημαντικά γιατί είναι σημαντικό εργαλείο μόχλευσης ε, και έχουν συγκεντρώσει πάνω από 8 δισεκατομμύρια ε, ευρώ για ε, μετοχές δάνεια και εγγύησεις. Είναι σημαντική λοιπόν αυτή η υποστήριξη όπως καταλαβαίνετε των ταμείων και της συνοχής γενικά στην οικονομία. Αυτό γίνεται ακόμα πιο εύγλωτο ε, στην επόμενη γραφική παράσταση ε, στο ρόλο που παίζει η πολιτική συνοχή για τις δημόσιες επενδύσεις. Βλέπετε ότι μισές περίπου χώρες, μισές περίπου επαναλαμβάνω χώρες, εποφελούνται από την πολιτική μας. πάνω από 30% των δημοσίων επενδύσεων και μπορεί να φτάσει αυτό και μέχρι το 70 και για ορισμένες χώρες και ακόμα παραπάνω. Ιδιαίτερα για την Ουγγαρία πάνω από 90%. Τα στοιχεία αυτά και τα δεδομένα δεν αντανακλούν καν το ότι γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο, γιατί πολύ συχνά Μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλη σημασία σε εθνικό επίπεδο, αλλά σε περιφερειακό επίπεδο πολύ συχνά τα δικά μας κονδύλια είναι η μόνη δυνατότητα των περιφερειών να υποστηρίξουν ουσιαστικά τις επενδύσεις, ιδιαίτερα σε καιρούς κρίσης. Τώρα, πώς ανταποκριθήκαμε στην κρίση. Ξέρετε ότι τα προγράμματα είχαν σχεδιαστεί πριν από την κρίση και χρειάστηκε να τα προσαρμόσουμε στις νέες προκλήσεις. Πρόκληση πρώτη. Η εθνική και οι περιφερειακοί προπολογισμοί γνώρισαν τεράστια συμπίεση για εξυγίανσή τους, δηλαδή η εθνική συγχρηματοδότηση απειλεί το. Και τι έπρεπε εμείς να κάνουμε, να αντιδράσουμε και να αυξήσουμε την κοινοτική συγχρηματοδότηση, πράγμα που κάναμε. Και ξέρετε ότι αυξήσαμε τις προκαταβολές το 2009 πάνω από 6,2 δις εκατομμύρια. Επίσης ε, το ποσοστό συγχρηματοδότησης ε, φτάσαμε στην οροφή ε, πάνω από 28 δισεκατομμύρια και για τις χώρες που είναι σε μνημόνια, σε προγράμματα, αυξήσαμε ακόμα περισσότερο τη συγχρηματοδότησή μας. Και έτσι βρέθηκαν άλλα 1,8 δισεκατομμύρια. That, Λοιπόν, τι βλέπουμε, ότι χρειάστηκε να αλλάξουν τα ποσοστά οι συντελεστέ σε χρηματοδότηση αλλά και να προσαρμοστούν τα προγράμματα στα νέα δεδομένα και στις νέες ανάγκες. Δηλαδή, χρειάστηκε ανακατανομή των κονδυλίων σε μεγάλο βαθμό πάνω από 45 δισεκατομμύρια, 13% δηλαδή. Είναι σημαντικό αυτό το ποσό και σαφές γιατί πολλά από τα προγράμματα δεν ήταν σχεδιασμένα ε, ώστε να καλύπτουν τις νέες ανάγκες, ε, οι οποίες είναι η ανεργία των νέων και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως γνωρίζετε, έχουμε τις περίφημες ομάδες δράσης το 2012 και συνολικά οι δράσεις αυτές βοήθησαν ένα εκατομμύριο νέους και 50.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. καθώς ε, μειωνόταν η οικονομία, μειωνόταν και η οικονομική δραστηριότητα και δεν μπορούσε να επεκταθεί η καινοτομία, γι' αυτό χρειάστηκε να προσαρμοστεί και η επιλεξιμότητα και αυξήθηκε στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στην κοινωνική στέγη και σε άλλους τομείς για να διευκολύνουμε την κατάσταση επιτόπου με απλουστευμένες επιλογές για το κόστος, ε, Πολλές φορές εμείς αποζημιώναμε ε, τα μεγάλα προγράμματα ακόμα πριν ληφθεί η απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να απλουστεύσουν και από πλευρά τους τις διαδικασίες. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν πολλές χώρες που επιβάλλουν επιπλέον κανόνες στους δικούς μας. Ε, Χρυσών, το λεγόμενο gold plating. Λοιπόν, εδώ τώρα τι βλέπουμε στην επόμενη γραφική παράσταση. Πόσο με την αυξημένη ροή των κοινοτικών κονδυλίων οι εθνικές ανάγκες συγχρηματοδότησης μειώθηκαν. Αυτό είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό για χώρες όπως η Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία και Λετωνία. Πάνω από 40% είναι η μείωση της εθνικής συγχρηματοδότησης και την Ιταλία πάνω από 20%, την Ισπανία, τη Λιθουανία και τη Ρουμανία αντίστοιχα. Περίπου 20% για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ τώρα βλέπετε την ανακατανομή, τον αναπρογραμματισμό των κονδυλίων και βλέπετε ότι ε, συνολικά, όπως σας είπα, ήταν 13%. Μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία και διαφορά μεταξύ των κρατών μέλων. Δεν θα σας εκπλήξει ότι ιδιαίτερα χώρες που έχουν μνημόνια ε, προγράμματα ξεπέρασαν το 20% αρκετά. Αυτά λοιπόν ως ε, περιγραφή τι έγινε με την κρίση και με τα διάφορα κράτη-μέλη που πλήττονται από τέτοια μέτρα. Τώρα, έρχομαι στην απορροφητικότητα των κονδυλίων. Αυτή η γραφική παράσταση σας δείχνει τις ε, προσωρινές πληρωμές της ενδιάμεσης μέχρι τα τέλη του 2013. Τι σημαίνει αυτό, όχι τις προκαταβολές. Όχι μόνο αυτές που έχουμε καταβάλει, αλλά αυτές που έχουν προγραμματιστεί αλλά δεν εξοφλήθηκαν για διάφορους λόγους. Και μεταξύ άλλων, όπως γνωρίζετε, διότι το ταμείο ήταν μείον στα τέλη του περασμένου έτους. Ποια είναι όμως τα ευχάριστα νέα τώρα. 60% απορροφητικότητα συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθόλου ευκαταφρόνιστο, πολύ αξιοσέβαστο αυτό το στοιχείο, αλλά δείχνει ότι παρόλα αυτά μας μένει 40% να καλύψουμε. Για το 2014 και 2015 πρέπει να πούμε ότι θα είναι χρόνια με πάρα πολύ δουλειά. Επίσης διαπιστώνεται ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά από χώρα σε χώρα. Δηλαδή, έχουμε ιδιαίτερα χαμηλή απορροφητικότητα στη Ρουμανία, Βουλγαρία, Σλοβακία, Μάλτα, Ιταλία, Ουγγαρία και Τσεχική Δημοκρατία. Βλέπετε εδώ στα αριστερά της γραφικής παράστασης της χώρας αυτής. Γίνονται πολλές προσπάθειες σε αυτές τις χώρες για να βελτιωθεί η κατάσταση και εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους βοηθήσουμε. Στη συνέχεια θα επεκταθώ λίγο παραπάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά πριν έρθω σε αυτό να πούμε δύο λόγια για την οικονομική διαχείριση. Άλλο κρίσιμο θέμα για την ε, απορρόφηση των κονδυλίων και την εκτέλεση. Θα πρέπει να βεβαιωνόμαστε πάντα ότι είναι ε, σωστές οι δαπάνες, νόμιμες. Αυτό είναι πάρα πολύ επίκαιρο γιατί γίνεται η συζήτηση για την απαλλαγή και την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Είναι κρίσιμο και από πλευρά τη αξιοπιστία τη πολιτική μα. Δεν θα πρέπει να είμαστε εδώ σε αμυντική θέση, στάση, διότι έχουμε δημιουργήσει δομές πάρα πολύ ισχυρέ και για τη διαχείριση και για τον έλεγχο το σύστημά μας. Και γενικά οι διαχειριστικέ αρχές, οι ελεκτικές ε, ε, αρχές και όλοι οι ενδιαφερόμενοι ε, εργάζονται πάρα πολύ σκληρά. Βεβαίω το ξέρω ότι χωράνε βελτιώσεις, αλλά δεν πρέπει να παίρνουμε μια αμυντική στάση, να βελτιωθούμε μπορούμε πάντα. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε λοιπόν μια διπλή προσέγγιση, ε, προληπτική και διορθωτική. Ποια είναι η προληπτική. Προσπαθούμε να αποφεύγουμε ατασταλίες, ε, παρατυπίες, αλλά σε περίπτωση που συμβαίνουν θα πρέπει να διορθώνονται. Και όπως γνωρίζετε, αυτό καταρχάς και καταρχήν είναι ευθύνη των κρατών μελών σας ανέφερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε μια εποπτική ευθύνη και όχι μόνο. Έχουμε ε, μπει και εμπλακεί και σε πολλές προληπτικές δράσεις με κατευθυντήριες γραμμές. Πάνω από 50 σημειώματα έχουμε. Ε, κάνουμε σεμινάρια, κάνουμε ενημερώσεις. Πρόσφατα για τη λήξη, του κλείσιμο της περίοδου 2007-2013 και κατά τις αποστολές ελέγχου οικονομικού ε, θέτουμε αυτά τα ζητήματα υπόψη των ενδιαφερομένων και στις αιτήσεις συνεδριάσεις που κάνουμε. Και από πλευράς ε, καθοδήγησης και πρόληψης κάνουμε πολλά και στο μέλλον ακόμα περισσότερο όπως θα σας εξηγήσω αργότερα. Άλλο ε, προληπτικό μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας είναι το εξής. Οπότε βλέπουμε ανεπάρκειες στη διαχείριση και στην εκτέλεση κάποιου προγράμματος, προειδοποιούμε την αρμόδια αρχή ότι θα πρέπει να διορθώσει αυτά τα στρεβλά και τα κακό σκήμενα. Και για να αποφύγουμε την καταβολή πληρωμών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αχρεωστήτως καταβληθέν ποσών, προειδοποιούμε τα κράτη-μέλη να μην κάνουν τις πληρωμές τους. Αν το κάνουν, δικαίωμά τους είναι στο κάτω-κάτω. Και καμιά φορά κάνει και καλό στα τέλη του έτους. Αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να διακόπτουμε και να αναστέλουμε τις πληρωμές μας, εάν δεν διορθωθεί εγκαίρως ε, αυτή η παρατυπία. Και Ξαναρχίζουμε τις πληρωμές μόνο εφόσον έχουν διορθωθεί ε, αυτές οι καταστάσεις και έχουμε και τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να επαναληφθούν στο επόμενο διάστημα ή στο μέλλον. Πάνω από 100 ήταν οι περιπτώσεις που διακόψαμε τις πληρωμές το 2013 και το συνολικό ποσό ήταν περίπου 4 δισεκατομμύρια. Και έχουμε και ψηλό ε, ποσό στις διορθώσεις. Ένα δισεκατομμύριο για όλες τις περιπτώσεις του 2013. Επόμενη διαφάνεια. Δείχνει πόσο σοβαρά παίρνουμε αυτά τα θέματα. Είναι σημαντικό αυτό το εργαλείο της πρόληψης για να μειωθεί το ποσοστό των σφαλμάτων. Βλέπετε εδώ σε πόσες περιπτώσεις διακόψαμε και αναστήλαμε τις πληρωμές, έχουν αυξηθεί αυτές κατά τη διάρκεια των ετών και επίσης τα ποσά έχουν αυξηθεί. Πολλά σας είπα τώρα για πολλά διαδικαστικά, αλλά έχει σημασία να δούμε και στην ουσία ε, τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά, από τις ατασταλίες, τις παρατυπίες και πού συμβαίνουν αυτά κατά κύριο λόγο ε, και θα πρέπει να δούμε τι λέει και το ελεκτικό συνέδριο σχετικά ποιες είναι οι ε, βασικές, τα βασικά είδη σφαλμάτων. Βλέπετε εδώ πέρα ότι έχουμε τις δημόσιες συμβάσεις που αντιστοιχούν στο 50 περίπου της 100 των σφαλμάτων. Και έπειτα έχουμε και το ζήτημα της επιλεξιμότητας που αντιστοιχεί και αυτό σε πολύ μεγάλο ποσοστό μη επιλεξιμότητα προκειμένου. Και αυτό βέβαια με τη σειρά του αποτελεί πρόβλημα. Και ουσιαστικά, αν λάβετε αυτά τα δύο στοιχεία μαζί, έχετε τα τρία τέταρτα των συνολικών σφαλμάτων που εντοπίζουμε. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι το ότι επικεντρωνόμαστε σε αυτούς τους δύο τομείς σφαλμάτων, δημόσιες συμβάσεις και επιλεξιμότητα. που είναι και ένα γενικότερο πρόβλημα, ιδίω στις διοικήσεις εκείνες που δεν έχουν την απαραίτητη ικανότητα να αξιολογούν τις διάφορες δαπάνες που μπορούν να υποστηριχθούν, να δικαιολογηθούν. Θέλουμε όμως να επεκτείνουμε κάπως το πεδίο αυτό και να μην επικεντρωνόμαστε μόνο σε έναν τομέα, γιατί αυτό το οποίο διακυβεύεται είναι η ίδια ικανότητα απορρόφησης από τα κράτη-μέλη και αυτό με τη σειρά του συνδέεται με την διοικητική ετοιμότητα και ικανότητα αυτών των κρατών. Και αυτό το βλέπετε ξεκάθαρα στην επόμενη γραφική παράσταση. Βλέπετε εδώ πέρα ότι έχουμε προσπαθήσει να δημιουργήσουμε μια γραφική παράσταση με δύο βασικούς άξονες. Στον άξονα έχουμε το επίπεδο απορρόφησης και στον άλλον την, ένα ποσοστό, έναν δίκτυ διοικητική ικανότητα. Βασιζόμαστε εδώ πέρα σε έναν δίκτυ διακυβέρνηση τη Παγκόσμια Τράπεζα. Αυτό το οποίο βλέπουμε ξεκάθαρα είναι ότι σε περίπτωση αδύναμης ε, διακυβέρνησης έχουμε και χαμηλή απορροφητικότητα, ενώ σε επίπεδο ισχυρής διακυβέρνησης και διοικητικής ικανότητας έχουμε και υψηλά επίπεδα απορρόφησης. Ουσιαστικά, όσο καλύτερη η διακυβέρνηση, τόσο καλύτερα και τα επίπεδα απορρόφησης. Και γι' αυτό το λόγο, την τελευταία φορά που να διοργανώσαμε τη Γενική Διεύθυνση Regio, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μία νέα αρμοδιότητα, η οποία επικεντρώνεται ακριβώς αυτό, διοικητική ικανότητα. Ακριβώς επειδή θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα για το τομέα αυτό, προκειμένου να είμαστε σε θέση να δώσουμε τις απαραίτητες ε, συμβουλές και την απαραίτητη καθοδήγηση στα κράτη-μέλη, προκειμένου να βελτιώσουν τη διοικητική τους ικανότητα και να, καταφέρουν να, γίνουν, να καταφέρουμε να κάνουμε και εμείς τις απαραίτητες διορθώσεις. Στην τελευταία αυτή διαφάνεια βλέπετε τις συγκεκριμένες αυτές δράσεις που εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε αποφασίσει να αναλάβουμε για να αυξήσουμε τη διοικητική ικανότητα των κρατών μελών, καθότι ένα βασικό πρόβλημα, όπως είδατε, είναι οι δημόσιες συμβάσεις. Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο δράσης για τις δημόσιες συμβάσεις, όχι μόνοι μας, η Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο δηλαδή, αλλά και σε συνεργασία και με άλλε Γενικέ Διευθύνσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα με τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερική Αγορά, DG Markt. Νομίζω ότι ουδέποτε είχαμε μια τόσο έντονη διυπηρεσιακή συνεργασία στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι το έργο το οποίο κάνουν οι μεμονωμένε Γενικέ Διευθύνσει θα είναι πλέον συντονισμένο και επί του παρόντος επικεντρωνόμαστε περισσότερο στην μακροοικονομική αιρεσιμότητα στα νέα προγράμματα, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι η εξάντε μακροοικονομική αιρεσιμότητα θα τηρείται και αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, να γνωρίζουμε ποιες θα πρέπει να είναι οι δράσεις που θα αναλυφθούν. Λέμε επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη καθοδήγηση για τους συμμετέχοντες στις δημόσιες συμβάσεις και θα έχουμε γι' αυτό τις συμβουλές, την ε, εμπλοκή κάποιων εμπειρογνωμόνων. Κατά αυτόν τον τρόπο ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε τον τομέα αυτό των δημοσίων συμβάσεων και ο έλεγχος θα γίνει καλύτερος. Το επόμενο σχέδιο το οποίο έχουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα κοινό σύστημα ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης, τεχνογνωσίας για το πώς μπορούμε να χειριστούμε τα ταμεία της πολιτικής συνοχής. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές ε, οι εμπειρογνώμονες και οι γνώστους τελικά βρίσκεται πολύ μακριά και είναι αποκομμένοι από το τοπικό περιφερειακό επίπεδο, εκεί που πραγματικά δηλαδή τους χρειαζόμαστε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης στο Μάστριχτ να διερευνήσουμε περισσότερο την πτυχή της ζήτησης και την πτυχή της προσφοράς και να δούμε τελικά πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καλό σύστημα ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων Ήδη γνωρίζουμε ότι άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες στο παρελθόν έχουν λειτουργήσει καλά, μπορούμε λοιπόν να εμπνευστούμε από αυτές, αλλά θέλουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε ένα μέσο το οποίο είναι προσαρμοσμένο σε ανάγκες της πολιτικής συνοχής. Πέρα όμως από τις δράσεις για τις ε, δημόσιες συμβάσεις αποφασίσαμε να διοργανώσουμε και κάποια εξειδικευμένα σεμινάρια, εργαστήρια στα κράτη-μέλη για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς. Ε, για πρώτη φορά το Δεκέμβριο στις Βρυξέλλες διοργανώσαμε ένα τέτοιο σεμινάριο για την καταπολέμηση της ε, διαφθοράς στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων και είχαμε μάλιστα και τη συνεισφορά της Transparency International, της Διεθνούς Διαφάνειας. Θα δώσουμε συνέχεια τώρα στην πρωτοβουλία αυτή και θα δημιουργηθούν, όπως σας είπα, εξειδικευμένα εργαστήρια σε διάφορες χώρες, όχι μόνο για να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση για το πρόβλημα αυτό, της διαφθοράς και της απάτης δηλαδή, αλλά και για να παρουσιάσουμε συγκεκριμένα μέσα καταπολέμησης των φαινομένων αυτών. Για παράδειγμα, υπάρχουν κάποια τα λεγόμενα σύμφωνα ακεραιότητος προκειμένου να καταπολεμήσουμε πιο αποτελεσματικά την διαφθορά και την απάτη στις δημόσιες συμβάσει. Και τέλος, για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, ξέρετε ότι για αυτήν προβλέπονται σημαντικές θεμελιώδεις αλλαγές και έχουμε ένα, προβλέπουμε ένα στοχευμένο πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο θα είναι ανοιχτό για όλους εμπλεκόμενους στα κράτη-μέλη, ωστόσο θα πρέπει να είναι στοχευμένο κυρίως για τις χώρες εκείνες που έχουν χαμηλή διοικητική ικανότητα. Θέλουμε λοιπόν κάποιες μικρότερες εξειδικευμένες ομάδες, 30 περίπου ατόμων, προκειμένου το πρόγραμμα αυτό κατάρτισης να είναι όντως αποτελεσματικό. Κυρία Πρόεδρε, πολύ συνοπτικά αυτά είχα να σας πω. Προσβλέπω στη συζήτηση που θα ακολουθήσει και όπως βλέπετε εμείς πολύ ενεργά παρακολουθούμε την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής επιτόπου και προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τη βοήθεια των κρατών μελών το πρόγραμμα αυτό, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και κάνουμε όλο και περισσότερα πράγματα όπως βλέπετε στο προληπτικό αυτό τμήμα προκειμένου να βοηθήσουμε τελικά τα κράτη-μέλη να διαχειρίζονται διοικητικά καλύτερα τα διαφορετικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχή. Κατά αυτόν τον τρόπο πραγματικά συμβάλλουμε στο να δημιουργηθούν καλύτερε συνθήκε απασχόληση και οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε μπορείτε να μας υπενθυμίσετε τι θα γίνει με τις πληρωμές, τις ε, καταλεκτικές ημερομηνίε, πώς προβλέπονται όλα αυτά για το διάστημα μέχρι το 2014. Μιλώ υπό τον έλεγχο του συναδέλφου βεβαίως. Στην πράξη, οι πληρωμές πρέπει να έχουν καταβληθεί για το 2014 και 2015. Αυτή είναι η περίοδος επιλεξιμότητας. Αυτά μετράνε για την ε, υλοποίηση στην πράξη. Προκειμένου να υπάρξουν αξιώσεις, ε, ενδιάμεσες αξιώσεις προς την Επιτροπή και τα τελικά έγγραφα χρειάζεται νομίζω περισσότερος χρόνος. Υπάρχουν, ε, διατίθονται 18 μήνες νομίζω. Μάρτιος του 2017 είναι η ημερομηνία. Αλλά αυτό που πραγματικά μετράει είναι το 2014 και το 2015, στην πράξη. Διότι μετά έχει κλείσει το θέμα. Είναι περισσότερο διοικητική η δουλειά που μένει. Για να ετοιμαστούν οι τελευταίες αξιώσεις πληρωμών και οι απαραίτητες εκθέσεις για το κλείσιμο των λογαριασμών. Ευχαριστούμε κύριο Γκουλμάνης. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσει. Για το κύριο Γενικό Διευθυντή. Πρώτον, πώς παρακολουθείτε τους αριθμούς για τις πρόσθετες πληρωμές. Διότι αν δούμε την παρουσίασή σας, βλέπουμε για τις επενδύσεις να υπάρχει ένας πίνακας με 95% για την Ουγγαρία, με μεγάλο ποσοστό δημόσιων επενδύσεων. Το 95% δηλαδή είναι κονδύλια ευρωπαϊκής συνοχής μαζί με εθνική συγχρηματοδότηση. Όμως αν είναι 95% για την Ουγγαρία δεν ε, πληρούν τις συνθήκες επιλεξιμότητάς τους. Δεν είναι όμως η μόνη χώρα, είναι και η Λιθουανία και η Σλοβακία που δεν τα πάνε τόσο άσχημα. Τι σημαίνει αυτό το 2010 υπήρξε ένα έγγραφο επαλήθευσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκεί λεγόταν ότι όλες οι χώρες πέραν των κονδυλίων που παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση από την πολιτική συνοχή πρέπει να προβλέψουν και πρόσθετη χρηματοδότηση από τα, από το κρατικά δημοσιονομικά, από τον κρατικό προπολογισμό. Αυτό το δέχεστε. 94 δις ευρώ ήταν αυτά σε μια πρώτη φάση. Εάν το διαιρέσετε δια του 336 που αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μεγάλο ποσό, είναι κάτι λιγότερο από το 1 τρίτο. Τι έγινε τελικώς. Εσείς θεωρήσατε ότι λόγω της κρίσης μπορούν οι χώρες να πάνε από τα 94 ε, δις στα 80, δηλαδή 40,9% το 2010 ε, μείωση. Πώς θα παρακολουθήσετε τους αριθμούς αυτούς της, των πρόσθετων κοντιλίων θα επιτρέψετε σε κάποιες χώρες λόγω των προβλημάτων των κρατικών τους δημοσιονομικών και του προπολογισμού τους να κατέβουν κι άλλο, να μειώσουν κι άλλο τα ποσοστά συγχρηματοδότησης. Γιατί ο πρώτος σας πίνακας δείχνει ότι οι χώρες δεν πληρώνουν τις ε, προϋποθέσεις που τους έχουν τεθεί. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό λοιπόν. Αυτό είναι η πρώτη, η πρώτη μου ερώτηση, εάν ήμουν σαφής. Το δεύτερο αφορά αυτό που είπατε για τους λόγους καθυστέρησης ε, των ε, της απορρόφησης κονδυλίων. Το 75% είπατε ότι είναι η επιλεξιμότητα και οι ε, δημόσιοι διαγωνισμοί. Όμως είδαμε και κάποιες αξιώσεις πληρωμών να αναστέλλονται και επίσης αριθμούς από την κρίση ένα έτος. Εάν ισχύει αυτό με τις δημόσιες προμήθειες που είπατε, πώς το εξηγείτε ότι η ανάπτυξη συνεχίζεται ε, το τελευταίο διάστημα αυτής της περίοδου 2012-2013 και εφόσον υπάρχουν καθαστηρήσει. Διότι εφόσον κάποιο ξεκινήσει ένα πρόγραμμα, πρέπει να έχει κάνει και ένα δημόσιο διαγωνισμό προηγουμένω, σωστά. Και μόνον μετά, διότι το 2013 δεν έχουμε νέα προγράμματα, και μετά με την καθυστέρηση διορθώνεται η κατάσταση και έτσι αρχίζετε εσεί να μετράτε το πώ αυξάνονται οι καθυστερήσεις οι διακοπές οι αναστολές από τη δική σα πλευρά. Βεβαίω, κάθε χώρα έχει δικό τους, δικό δική τη νομοθεσία για τι δημόσιε προμήθειε. Δεν υπάρχει ένα μόνο νόμο για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημα λοιπόν είναι, τι θα κάνετε από εδώ και στο εξή. Τι θα κάνετε αφού κάθε χώρα έχει τη δική τη νομοθεσία. Και ποια θα είναι η δική σα τοποθέτηση. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Γιατί η Λιθουανία είναι υπαριθμόν ένα στην απορρόφηση και του Ταμείου Συνοχής και των Διευθυντικών στο 2013. Είναι διαφορετική κατάσταση εκεί. Αντιστρέφουν τη σειρά των δημόσιων προμηθειών. Αρχικά η ανοιχτοί διαγωνισμοί και το σύστημα ανοιχτών διαγωνισμών ισχύει και μετά μόλις ο δικαιούχος ε, πληρώσει όλες τις προϋποθέσεις τότε φέρνουν ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι διαφορετικό από τις άλλες χώρες. Πρώτα είναι κανείς επιλέγεται για ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά μετά άμα δεν ε, συμφωνεί με τους ε, κανόνες του εθνικού νόμου για τους δημόσιους διαγωνισμούς, απορρίπτεται. Πάντως για την ε, επιλογή και τα προσόντα ε, είσαστε πολύ αισιόδοξου μιλήσατε για τη σχετική ε, διακυβέρνηση και απορρόφηση. Εάν δείτε ότι ο συσχετισμό είναι μόλις 20%, 7 χώρες από τις 27 δείχνουν ότι επιβεβαιώνουν αυτό το συσχετισμό. 25% με συγχωρείτε, αλλά το 20% δείχνουν ότι έχουν ισχυρή διακυβέρνηση με καλή απορρόφηση, αλλά υπάρχουν και άλλοι τόσοι που έχουν χαμηλή διακυβέρνηση και υψηλή απορρόφηση. Δεν είναι 100% λοιπόν σωστός αυτός ο σχετισμός που αναφέρατε. Εάν δείτε τον αριθμό όλων των χωρών, αυτό λοιπόν με απασχολεί εμένα. Δεν είναι 100% σωστός ο σχετισμός. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσέλερ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, στα πολωνικά και στα γερμανικά, κύριε Ντέφα, για τη συλλογική ανάλυση, την τόσο εξαντλητική ε, και τόσο νυφάλια, ε, αλλά καμιά φορά είναι και αφυπνιστική, για να το πω έτσι. Εγώ είμαι ακρεφνής υποστηρικτής ε, της περιφερειακής πολιτικής, της διαθωτικής και της συνοχής που να συνδέεται με την περιφερειακή πολιτική. Είμαι ένθερμος υποστηρικτής όλων αυτών. Τι ζούμε όμως αυτόν τον καιρό. Τα επενδυτικά ταμεία που είναι σε περιφερειακό επίπεδο πολλές φορές η μοναδική ε, δυνατότητα επενδύσεων, από ό,τι φαίνεται ε, συγκεντρώνονται στα κράτη Ακόμα και κράτη με περιφερειακό, με ομοσπονδιακό χαρακτήρα, που δεν πρόκειται για τη Γερμανία εδώ, ε, τα συγκεντρώνουν σε κεντρικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο πρώτα και οι περιφέρειες όλο και περισσότερο εξαρτώνται από αυτό που αποφασίζεται για λογαριασμό τους σε κεντρικό εθνικό επίπεδο. Δεν έχει πολύ μεγάλη σχέση πια αυτό με περιφερειακή πολιτική όμως. Αυτό μπορεί για μικρότερες χώρες να είναι εντάξει και να έχει νόημα ε, για χώρες που έχουν, ξέρω εγώ, ένα-ενάμιση εκατομμύριο κατοίκους, να μην υπάρχει κατακαιρματισμός, αλλά όταν είναι μεγαλύτερα τα κράτη, ε, παίζει ρόλο και η περιφερειακή διάσταση και υπάρχουν και περιφερειακές διαφορές. Θα πρέπει να διατηρηθεί αυτή η περιφερειακή διάσταση. Κάτι άλλο που θεωρώ επίσης ε, σοβαρό και κρίσιμο γιατί έχουμε μπει σε προεκλογική σχεδόν εξατία, είμαστε παραμονές εκλογών και τα ευρωπαϊκά θέματα ε, έρχονται περισσότερο στο προσκήνιο και στις χώρες μας στην κοινή γνώμη από ό,τι γενικότερα. Και το θέμα είναι οι διάφορες αξιώσεις που έχουμε και οι διάφορες δυνατότητες που παρέχουμε εάν συμπίπτουν με την πραγματικότητα. Είπατε ότι είναι πάνω από 900 τα χρηματοδοτικά μέσα που χρησιμοποιούνται για χώρες, περιφέρειες κτλ για τους ανθρώπους που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες κοινωνικές. Αυτά πώς πανώνται; Μετά από πρωτοβουλία της δικής μας Προέδρου, πριν από δύο-δυόμιση χρόνια αν δεν απατώμε, αποφασίσαμε και για ένα μέσο ε, διαμερισμού ε, και του ρίσκου και του κινδύνου. Δηλαδή σε χώρες όπου έχει καταρρεύσει ο τραπεζικός τομέας ή που έχει δυσκολίες ε, να μπορέσουν να συνεχίζονται τα προγράμματα. Έκανα μια ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πόσες χώρες είναι αυτές ε, που είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτό το μέσο και ποιες το ε, αξιοποίησαν. Κανένας, καμία χώρα δεν το ζήτησε καν. Και τι γίνεται με τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά μέσα που διαθέτουμε στα κράτη-μέλη. Άλλη επίκαιρη συζήτηση που γίνεται. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή στρατηγική για τους Ρωμά αναπτύξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ στην Επιτροπή μας έχουμε τη δυνατότητα διαρθρωτικά κονδύλια να πηγαίνουν στην ένταξη και στην βελτίωση ε, της διαβίωσης κοινωνικά περιθωριοποιημένων ομάδων που δεν είναι η Ρωμά αλλά κυρίως η Ρωμά ε, μόνο. Ε, από ό,τι φαίνεται σε εθνικό επίπεδο είναι μάλλον περιορισμένες οι επιτυχίες. Αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε γιατί καθορίζουν τη συζήτηση. Εμείς αποφασίζουμε ε, οδηγίες για την αποτελεσματικότητα της ενέργειας με πολύ υψηλές αξιώσεις και ακόμα και την περασμένη εβδομάδα το Κοινοβούλιο έκανε πιο αυστηρούς τους στόχους με τις εξής επιπτώσεις, ας πούμε την κοινωνική στέγη κοινωνικές κατοικίες ή ενίκαιο ε, που να μπορεί να το πληρώνει ο μέσος ε, δικαιούχος. Αυτά είναι αντιπαραγωγικά που αποφασίζουμε. Στη Βερολίνο ε, χρειαζόμαστε νέα στέγη, αλλά υπάρχουν εταιρείε κατασκευαστικές όπου είναι 6,5 ευρώ για το τετραγωνικό η τιμή ε, ε, χωρίς ακόμα να υπολογίζει τη φέρμανση κτλ. Ε, είναι αυτό οροφή. Μα για το Βερολίνο δεν είναι τιμές αυτές και μας το λένε οι κατασκευαστές, οι εργολάβοι. Υπάρχουν όλα αυτά τα μέτρα που ακόμα και αν τους δώσουν δωρεάν το οικόπεδο, δεν μπορούν να χτίσουν με κόστος κάτω από 10 ευρώ το τετραγωνικό. Και επίσης μπαίνει και το θέμα των κρατικών ενισχύσεων, αν ενισχυθούν από το κράτος, ε, μπαίνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού και φωνάζει ότι τι είναι, αυτά, τι είναι αυτές οι κρατικές ενισχύσεις που υποστηρίζουν την ανέγερση κατοικιών. Ε, υπάρχει λοιπόν μια ολόκληρη πλειάδα θεμάτων όπου ήδη διαπιστώνουμε ότι τα μέσα και οι δυνατότητες δεν συμπίπτουν με την πραγματικότητα και με τον τρόπο που υλοποιούνται. Και είναι εύγλωτοι και οι αριθμοί η Επιτροπή Ελέγχου ε, του προεπολογισμού ε, θα τονίζει αυτά τα θέματα. Εγώ ε, όταν ήμουν ε, επικεφαλής σε ένα διαμέρισμα δημοτικό ε, είχα ξεχωριστή μονάδα για την προκήρυξη διαγωνισμών με, ε, με πολλούς υπαλλήλους και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Τώρα αυτό θεωρείται πολυτέλεια και απολύουν και δημοτικούς εργαζομένους. Δηλαδή πριν κάνει κανείς κάποιο σφάλμα για το οποίο σε καθίζουν στο εδόλιο θα πρέπει να δει τι δυνατότητες υπάρχουν στην πόλη μου το Βερολίνο έχουμε τώρα μια μεγάλη συζήτηση για ποιο λόγο είναι πολλά τα εκατομμύρια ε, από τα κονδύλια και κοινοτικά και ε, κρατικά που μας δίνει η γερμανική κυβέρνηση δεν απορροφώνται. Ένας από τους λόγους ήταν ότι δεν έχουμε τους υπαλλήλους εκείνους που χρειαζόμαστε και έχουν τα προσόντα και την ειδίκευση για να προκυρήσουν αυτούς τους διαγωνισμούς. Λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα που κρύβονται και πολύ χρώμα και πολυδιάστατα που κρύβονται πίσω από αυτή την έκθεση και τώρα που μπαίνουμε στην προεκλογική εκστρατεία θα πρέπει με συνοχή, όπως λέμε πολύ ωραία, να τα αντιμετωπίζουμε. Τα γενικά και όριστα δεν βοηθούν. Χρειάζονται συνεργασίες, εγκάρσεις των διαφόρων επιτροπών και θέλω να απευθύνω μια έκκληση στη Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο να προσπαθήσει να έρθει σε επαφή και με άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να υπάρξει συντονισμός για αυτά τα θέματα και συνεργασία. Διότι δεν μας βοηθάει καθόλου από τη μια να έχουμε καλές προθέσεις και καλές απαιτήσει και ξέρουμε ότι το καλύτερο εχθρός του καλού και οι καλύτερες των προθέσεων ε, δεν βοηθούν αν δεν εφαρμόζονται όλα αυτά στην πράξη και πάνε στο βρόντο όλες οι προσπάθειες για την πολιτική συνοχή, για τη διαρθρωτική πολιτική και για όλους τους στόχους μας. Ευχαριστώ. Okay, um, mm, after these three... Μετά από αυτές τις τρεις ε, παρεμβάσεις, ίσως να κάνω και εγώ κάποια σχόλια. Η ρεσιμότητα είναι ένα... Η προσθετικότητα είναι ένα πολύ ε, θέμα. Μπορεί να μας παραπλανήσει. Με ευρωπαϊκά κονδύλια δεν πρέπει να υποκαταστήσουμε κάτι που τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να είχαν κάνει από μόνα τους. Όμως, ε, θεωρητικά κιόλα δεν είναι πολύ εύκολο να υποθέσει κανείς τι θα είχε γίνει αν δεν είχαν υπάρξει τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η οικονομική κατάσταση είναι πολύ σημαντική. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει κανείς να επικρίνει, να μας επικρίνει που έχουμε προσαρμόσει τη συγκριτική αξιολόγηση για να μπορούμε να αποτιμήσουμε και την ε, συγκρισιμότητα, την, ε, συγγνώμη, την Θα ξέρετε ότι σε περιφερειακό επίπεδο δεν είναι το ίδιο αυτό που θα μπορούσαν να είχαν κάνει τα κρατημέλη προ και μετά κρίση. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Ακόμη και όταν μιλάμε για την προσθετικότητα. Οπότε, εντάξει έχουμε θεωρητικούς αριθμούς, αλλά σε μια πραγματικότητα που στην ουσία δεν ισχύει. Και Όπου και να πάω, μου λένε ότι ένα από τα προβλήματα για την χαμηλή απορρόφηση είναι ακριβώς και η διάθεση της ε, εθνικής συγχρηματοδότησης. Δεν διατίθεται. Εάν το δείτε λοιπόν και αυτό, εντάξει έχετε δίκιο, εάν μειώσουμε το ποσό της εθνικής συγχρηματοδότησης σίγουρα ο όγκος των επενδύσεων θα περιοριστεί, θα συρρυκνωθεί. Από τους αριθμούς όμως βλέπουμε ότι ακόμη και με μικρότερο επενδυτικό όγκο οι οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν για τις προμήθειες, για τους ε, διαγωνισμούς. Σίγουρα υπάρχουν διαφορετικέ εθνικέ νομοθεσίε, όμω πρέπει να συμμορφώνονται και με τι ευρωπαϊκέ οδηγίε. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Όταν ε, απαντούμε παραβιάσει, όταν βλέπουμε λοιπόν να υπάρχουν παραβιάσει ή ατασταλίε, αυτό συνήθω δεν έχει να κάνει με τι ιδιαιτερότητε των εθνικών νομοθεσιών για τι δημόσιε προμήθειε. Αυτέ οι παραβιάσει και ατασταλίε έχουν να κάνουν με την παραβίαση βασικών αρχών των ευρωπαϊκών οδηγιών. Έχουμε λοιπόν ευρωπαϊκές οδηγίες και ελπίζουμε ότι θα κάνουν τα πράγματα κάπως απλούστερα. Αλλά δεν είναι σωστό όταν πει κανεί ότι υπάρχουν τελείως οριοθετημένα τοπία διαφορετικά και ξεχωριστά μεταξύ τους ό,τι αφορά τις δημόσιες προμήθειες. Υπάρχει και η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία κυριαρχεί στο τοπίο. Για το συσχετισμό Δεν ισχύει κατά 100% αυτή η εξίσωση. Δεν, δεν αντιλέγω, αλλά έχει μεγάλη σημασία. Φυσικά υπάρχουν ένα σωρό ιδιαιτερότητες και λεπτομέρειες που κάνουν τη μια χώρα να είναι πάνω ή κάτω από τον άξονα, από τη γραμμή, αλλά βλέπετε ότι τάση υπάρχει. Υπάρχει μια κεντρική γραμμή, ένας κεντρικός άξονας, οπότε έχει και ενοιολογικά κάποια σημασία. Διότι αυτού του είδους η δυνατότητα είναι καθοριστική για τη βελτίωση της απορροφητικότητας. Και βεβαίως ε, έχετε δίκιο να λέτε ότι υπάρχουν πολλά σημεία όπου θα μπορούσαν να προκαλέσουν απορίες. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι στο μέλλον θα πρέπει να φροντίσουμε να εφαρμόζεται με συνέπεια και συνοχή η η πολιτική. Και μπορώ να σας πω ότι επειδή ασχολούμαι πάνω από 20 χρόνια ε, με διάφορους τομείς ε, αυτής της πολιτικής, ότι ο συντονισμός και η συνεργασία των διαφόρων υπηρεσιών στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ουδέποτε υπήρξε τόσο στενή όσο σήμερα. Ουδέποτε αρχίζει γενομένης από το γεγονός ότι για τη νέα προγραμματική περίοδο με τη δική σας υποστήριξη Ε, καταλήξαμε στους περίφημους όρους και προϋποθέσεις εκ των προτέρων, εξάντε, δηλαδή επενδύονται τα χρήματα μόνο όταν υπάρχουν δεδομένες κάποιες προϋποθέσεις νομικές, διοικητικές και άλλες στο περιβάλλον, στην ενέργεια, στις μεταφορές κλπ. Για να μπορέσει κανείς να διαπιστώσει καν κατά πόσο το κράτος μέλος τηρεί και πληρεί αυτά τα κριτήρια χρειαζόμαστε και προς τα εκεί εργαζόμαστε και πολύ ε, στενά για τις υπόλοιπες γενικές διευθύνσεις. Ή ας δούμε αυτό το παράδειγμα Smart Specialization ή ευφυής ειδίκευση. Είναι πολύ σημαντικά αυτό και από τη σκοπιά της περιφερειακής πολιτικής για να τονωθεί η ε, καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα των ε, περιφερειών. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με του συναδέλφους του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου στη Σεβίλη έχουν ιδιαίτερη μονάδα, όπου πάνε οι πελάτες μας εντός εισαγωγικών για να ζητούν συμβουλές. Συνεργαζόμαστε. Δεν λέω ότι είναι όλα τέλεια, αλλά είναι ακριβώς αυτή η κατεύθυνση που θέλουμε να πάρουμε για να συνεργαστούμε περισσότερο. Δεν συμφωνώ απολύτως όταν λέτε ότι υπάρχει μια τάση προς εθνικοποίηση, συγκέντρωση κεντρική δηλαδή περισσότερο των πόρων. Θα πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό όταν θα έχουμε όλα τα προγράμματα που βρισκόμαστε. Κοιτάξτε την ίδια σας τη χώρα. Σίγουρα δεν μπορεί να γίνει λόγος για εθνικό πρόγραμμα. Μάλιστα έχουμε ένα λιγότερο εθνικό πρόγραμμα. Κοιτάξτε προς δυσμάς ε, στη Γαλλία ας πούμε. Τώρα λαμβάνουν οι περιφέρειες ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην περιφερειακή πολιτική, ισχυρότερο από ό,τι στο παρελθόν. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για γενική τάση συγκέντρωσης και μη το εξή. Εθνικό πρόγραμμα δεν σημαίνει αυτόματα ότι δεν συμμετέχουν οι περιφέρειες στην εκπόνησή του. Ιδιαίτερα στο νέο κανονισμό με τα ITI στα λεγόμενα έχουμε ε, τις δυνατότητες πλέον και τα μέσα ε, να έχουμε και λειτουργικούς χώρους ας πούμε στο σχεδιασμό σε περιφερειακό επίπεδο που να αναλαμβάνουν την ευθύνη και να ε, κάνουν κτήμα τους τα προγράμματα τα οποία εκπονούν και αναπτύσσουν ίδιες. Νομίζω αυτό θα πρέπει να το δούμε κάπως διαφορετικά. Για τα χρηματοδοτικά μέσα, όπως συνήθως υπάρχουν πράγματα που πηγαίνουν καλά και άλλα που πάνε στραβά ή λιγότερο καλά. Ε, εντοπίσατε κάποιες αδυναμίες, αλλά ακριβώς και αυτό είναι ένας τομέας όπου ο νέος κανονισμός έρχεται να επιβάλλει πολύ πιο αυστηρούς κανόνες. Προσωπικά είμαι πάρα πολύ πεπισμένος ότι στο μέλλον ε, θα τα ελέγχουμε καλύτερα. Το θέμα των Ρωμά, μεγάλο πρόβλημα. Και στη νέα προγραμματική περίοδο θα το αντιμετωπίσουμε όλους ιδιαίτερο. Στην παλιά περίοδο, τουλάχιστον σε δύο κράτη-μέλη, Ουγγαρία και Σλοβακία είχαμε ειδικά προγράμματα. Διαφορετικά υπάρχουν διάφορες δράσεις στα πλαίσια της ένταξής τους. Και τα ποσά είναι αρκετά μεγάλα που έχουν προγραμματιστεί, τα οποία όμως δεν εφαρμόζονται, δεν εκτελούνται πάντα σωστά. Έχετε δίκιο εκεί και θα πρέπει να ε, το προσέξουμε και στο μέλλον αυτό. Αυτά. Νομίζω πάντησα, έτσι δεν είναι. Ευχαριστούμε ο κύριος Όρμπλεφτ. Σας ευχαριστώ κύριε Διευθυντά για αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες. Πολύ χρήσιμο ήταν που στο πρώτο μέρος της συνεδρίασής μας είχαμε συζήτηση με τους εμπειρογνώμονες. Μίλησαν και εκείνοι για τον τρόπο που δαπανούνται τα κονδύλια και για τις δυνατότητες καλής διοίκησης και τη σχέση με την καλή απορρόφηση. Όμως δεν δόθηκε μια σαφής απάντηση για το λόγο εξαιτία του οποίου σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχει υψηλή απορροφητικότητα αλλά ε, κακοδιοίκηση ενδεχομένω. Γιατί λοιπόν, γιατί σε κάποια κράτη-μέλη, στη δικό σας κατάλογο η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Τσεχία έχουν νομίζω τα χαμηλότερα ποσοστά στην ικανότητα απορρόφησης, στο ποσοστό απορρόφησης. Υπάρχει λοιπόν περίπτωση όχι να επωνυδίσουμε, αλλά τουλάχιστον να μας πείτε γιατί. Γιατί συμβαίνει αυτό. Υπάρχει θέμα διοίκησης ή υπάρχει κάποιο πρόβλημα ευρωπαϊκό, έξω ευρωπαϊκό. Είναι μια απλή ερώτηση πολιτικού χαρακτήρα, αλλά είναι σημαντικό για όλους μας. Και η δεύτερη ερώτηση που έχω είναι ότι αναφέρατε ότι το επίπεδο απορρόφησης είναι περίπου 60% σήμερα. Οπότε το 40% των ευρωπαϊκών κοντιλίων από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό χρειάζεται ήδη για το 14 και το 15. Εάν το συγκρίνουμε με τις ανάγκες των κρατών μελών, αυτές που μας αναφέρουν, θα πρέπει να έχουμε κονδύλια και το 14 και το 15 για να καλύψουμε όλες τις αξιώσεις που θα προκύψουν από την πολιτική συνοχή για αυτό το 40%. Ένα απλό συμπέρασμα, απλουστεύω κάπως τα πράγματα. Θα μπορούσαμε να πούμε στα κράτη-μέλη, παρακαλούμε, μη βιαστείτε. Μην βιαστείτε, γιατί αν ξεκινήσετε τα προγράμματα πολύ γρήγορα δεν θα υπάρχουν χρήματα. Και εντάξει, συζητάμε μετά το αν θα έχουμε εταιρικέ σχέσει, θα κρατήσει κάποιε μήνε η συζήτηση. Έναρξη των προγραμμάτων θα μπορούσε να γίνει το 2015. Οπότε οι πρώτες πληρωμές από το 2014 και το 2015 θα γίνουν το 2016. Αυτό είναι ένα πλουστευμένο συμπέρασμα. Όμω πολλέ φορέ οι άνθρωποι που εργάζονται στον ίδιο τον τομέα στην πράξη μα ρωτούν, ιδίω εμά του βουλευτέ, μα ρωτούν η μέθοδο για να ενισχυθεί ο έλεγχο και για να γίνονται οι αυτόματες διορθώσεις. Μήπως στόχο έχει να ε, εξοικονομήσει ε, κονδύλια από τον προπολογισμό. Δηλαδή, η πολιτική συνοχή και αυτή η μέθοδος που θα εφαρμοστεί στην πολιτική συνοχή, ίσω είναι ένα τρόπο για να μην δαπανηθούν πολλά χρήματα. Γιατί λένε ότι υπάρχουν προβλήματα. Ε, και έχουμε προβλήματα στα κενά του προπολογισμού, όχι μόνο για το 12 και το 2013, θα το έχουμε και το 2014 Μιλήσατε, φαντάζομαι γι' αυτό, και με τα εθνικά κοινοβούλια. Είναι λοιπόν ένα απλουστευμένο συμπερασμά ότι τα κράτη-μέλη τι μας λένε, γιατί μας ελέγχουν με τόσο απλοϊκό τρόπο ενώ όλο και πιο αυστηρή γίνεται η αρισιμότητα και μήπως προσπαθούν απλώς να κάνουν οικονομίες. Είναι πολιτικότατη και αυτή η ερώτηση. Παρακαλώ λοιπόν δώστε μου μια απάντηση διότι μας τη θέτουν την ερώτηση και καλούμαστε να δώσουμε απαντήσεις. Αυτές οι δύο, αυτά τα δύο επίπεδα, η δυνατότητα απορρόφησης και η υποστησιμότητα και η χάραξη πολιτικής είναι επίπεδα αλληλένδετα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα συνεχίσω να... θα μιλήσω σου ειδικά γιατί είναι η αυμένη μου γλώσσα. Έχω μια ερώτηση για τις δημόσιες προμήθειες. Πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα που δίνετε τέτοια προσοχή στις δημόσιες προμήθειες και το πρόγραμμα δράσης για, για τις δημόσιες προμήθειες. Είναι καλή, πολύ καλό πράγμα αυτό, διότι το να υπάρχει ανοιχτή και διαφανής διαδικασία για τους διαγωνισμούς στην πολιτική συνοχή είναι ίσως το καλύτερο μέσο για να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Ωστόσο, υπάρχει και ένας κινδύνος. Στα κράτη-μέλη, οι αρχές μπορεί να κατανοήσουν τον συσχετισμό μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ω ε, μια εντυγενέση περίπτωση διαφορά. Ένα παράδειγμα, είχαμε κάποια κλάστερ που ήταν πολύ επιτυχημένα, ε, κάποιες, ε, συνεργασίες για την καινοτομία, πολύ επιτυχημένες. Όλοι ωφελήθηκαν από την συνεργασία. Οι ιδιωτικέ, οι μικρέ ιδιωτικέ εταιρείε είχαν τη δική του πλατφόρμα, ήταν και υπεύθυνε για τα προγράμματα ίδιε. Αυτή η κοινή ανάληψη ευθύνη είναι καθοριστική για την επιτυχία. Όμω, εάν δεν υπάρχει αυτού του είδου η συνεργασία, δεν έχει κανεί δικαίωμα να λάβει κονδύλια από τα ταμεία. Εάν δεν υπάρξει συνεργασία δημόσιο-ιδιωτικού τομέα και συμμόρφωση με την Εθνική Νομοθεσία για τις δημόσιες Προμήθειες, δεν υπάρχει και η χρηματοδότηση. Οπότε όλοι είναι ε, πολύ καχύποπτοι για περιπτώσει διαφορά. Ευχαριστούμε, κυρία Μάλετιτ. Ευχαριστώ. Ε, είναι πολύ θετικά τα συμπεράσματα της μελέτης που παρουσιάσατε. Δείξατε ότι η απορρόφηση συσχετίζεται άμεσα με την καλή διακυβέρνηση και η καλή διακυβέρνηση συσχετίζεται αμεσά με τη διοικητική ικανότητα, την καλή διοίκηση. Χρειαζόμαστε ποιότητα και ποσότητα λοιπόν σε αυτούς που δουλεύουν στο σύστημα. Τώρα για τα μέσα, τα μέτρα μάλλον που σκοπεύετε να προτείνετε, που έχετε ήδη προτείνει στα κρατημέλη ώστε να τα προειδοποιήσετε να βελτιώσουν τις διοικητικές τους ικανότητες. Υπάρχει κάποια απλή έστω μεθοδολογία, κάποια μέθοδος που να δείχνει στα κάτι μελη πώς να διορθώσουν τις ε, διοικητικές τους πρακτικές και σε όλους τους τομείς που θα έπρεπε να καλύπτονται σε αυτές τις περιπτώσεις δίκησης. Επίσης, νομίζω ένα σημαντικό ε, στοιχείο για την ε, καλή υλοποίηση που θα θέλαμε να πετύχουμε, υψηλό επίπεδο δηλαδή απορρόφησης και χαμηλό επίπεδο ατασταλιών, είναι τα κονδύλια που θα μπορούσε να επενδύσει η κυβέρνηση σε προπαρασκευαστικές ε, φάσεις. Οι κυβερνήσεις δηλαδή δεν μπορούν απλώς να διασφαλίσουν, ούτε υποχρεώνται μόνο να διασφαλίσουν το σκέλος της ε, συγχρηματοδότησης, αλλά πρέπει να ε, είναι βέβαιες ότι θα δαπανώνται σωστά τα κονδύλια για την υλοποίηση του προγράμματος. 3 με 5% του συνόλου ε, της συνολικής αξίας ενός προγράμματος είναι η φάση της προπαρασκευής. Εάν θέλουμε να δαπανίσουμε λόγω χάρη ένα δις ευρώ, πρέπει να επενδύσουμε 300.000 εκατομμύρια 300 μάλλον εκατομμύρια για την προετοιμασία ενός προγράμματος. Ε, πρέπει λοιπόν οι κυβερνήσεις να αναλάβουν την ευθύνη για την παρακολούθηση αυτού του σκέλους και ε, σίγουρα περιορισμοί υπάρχουν, υπάρχουν και διαδικασίες ε, του υπερβολικού ελλείμματος, όμως υπάρχουν τρόποι στήριξης των κυβερνήσεων με διαφορετικά δημοσιονομικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν την καλή προπαρασκευή των προγραμμάτων που είναι και αυτή καθοριστική για την ε, καλή ε, λειτουργία της πολιτικής συνοχής. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανείς άλλος να θέλει το λόγο. Έχω και εγώ δύο σύντομες ερωτήσεις. Μετά από όσα μας είπε και ο Γιάννη, θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε για το ποια είναι αξία των αξιώσεων πληρωμών τις οποίες αυτή τη στιγμή εξετάζει η Γενική Διεύθυνση ε, Προπολισμών και που καλείται να πληρώσει. Και επίσης, Πότε θεωρείτε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν οι προκαταβολές. Πότε έρχεται η στιγμή από νομικής πλευράς που πρέπει να αρχίσετε να καταβάλλετε τις προκαταβολές. Θα υπάρξει πρόβλημα, θα είναι φέτος του χρόνου. Υπάρχει κάποια δυσκολία δεδομένων των όσων ισχύουν για τον προπολογισμό και το γεγονός ότι το Ευρωκοινοβούλιο δεν θα λειτουργεί για ένα διάστημα. Παρακαλώ. Uh, Θα ξεκινήσω με τις δικές σας ερωτήσεις, εκτέλους του προπολογισμού. Στο τέλος του έτους είχαμε 90 δισεκατομμύρια μεταξύ των διαφόρων περιφερειών όσον αφορά αιτήσει πληρωμών που είχαν γίνει και που εμείς δεν μπορούσαμε να καλύψουμε. Από αυτές, περίπου 4 περίπου δισεκατομμύρια διακόπησαν και ορισμένες αιτήσει πληρωμών ήρθαν ιδιαίτερα καθυστερημένα. Αν είχαμε αρκετά χρήματα, θα μπορούσαμε να είχαμε καταβάλει περίπου 10 με 11 δισεκατομμύρια. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν ήταν η διακοπή των πληρωμών τελικά αυτή η οποία ήταν ε, η πιο καθοριστική στη συγκεκριμένη περίπτωση. Στις αρχές βέβαια του έτους η δημοσιονομική κατάσταση είναι πάντα πιο προβληματική. Ελπίζω πάντως ότι από το απόθεμα του 2013 θα καταφέρουμε να καταβάλουμε 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2014. Αυτά μέσες άκρες είναι αυτά που μπορώ να σας πω στον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση για την εκτέλεση του προπολογισμού. Όσον αφορά τώρα τις προκαταβολές, αυτές θα καταβληθούν όταν εγκρίνουμε τα προγράμματα. και αυτό προβλέπεται κάποια στιγμή αργότερα το 2014. Πάντως, διαβεβαιώ την Επιτροπή σας ότι οτιδήποτε κάνουμε στα πλαίσια διαπραγματεύσεων, προτιμασίας, προγραμμάτων κτλ. δεν καθορίζεται από περιορισμούς στον προπολογισμό. Δεν καθορίζεται από μια κάποια στενότητα του προπολογισμού και απαντώ κατά αυτόν τον τρόπο στην ερώτηση του κυρίου Όλμπριχτ και νομίζω ότι σας έδωσε και κάποια αριθμητικά δεδομένα πριν από λίγο, τα οποία καταδεικνύουν ε, αυτό το πράγμα ξεκάθαρα. Και ας μην ξεχνάμε ότι η διακοπή των πληρωμών είναι απλώς μία διακοπή, μία προσωρινή αναστολή ουσιαστικά των πληρωμών, εφόσον βέβαια το κράτος μέλος αναλάβει τις απαραίτητες δράσεις. Στη συνέχεια τα χρήματα πάλι ξαναδίνονται στο κράτο μέλος, καταβάλλονται στη συνέχεια τα κονδύλια. Κάντε και κάποιες ερωτήσεις όσον αφορά την διοικητική ικανότητα. Ναι, εντοπίζουμε κάποια προβλήματα τα οποία πρέπει να διορθωθούν. Με την Τσεχική Δημοκρατία το 2011 ξεκινήσαμε ένα πολύ σημαντικό σχέδιο δράσης προκειμένου να βοηθήσουμε τις εκεί διοικητικές αρχές. Καταλαβαίνετε όμως ότι οι πρωτοβουλίες αυτές απαιτούν την πάροδο κάποιου χρόνου προκειμένου να έχουμε κάποιες θετικές επιπτώσεις. Και οι συνάδελφοι στην Τσεχική Δημοκρατία κατέβαλαν πολύ σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να καταφέρουν να βελτιώσουν και τη στρατηγική τους ικανότητα όσον αφορά την εφαρμογή των προγραμμάτων. Κύριε Νίλσον τώρα, δεν έχουμε εμεί κάποιο πρόβλημα με τα PPPs. Κάθε άλλο, θεωρώ ότι το μέσο αυτό είναι πολύ σημαντικό συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Είναι πολύ σημαντικές οι συμπράξεις αυτές και ξέρετε όταν οι κρατικοί, οι δημόσιοι προπολογισμοί είναι περιορισμένοι, προφανώς χρειαζόμαστε τα χρήματα του ιδιωτικού τομέα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο τροποποιούμε τη βάση συγχρηματοδότησης και λέμε ότι δεν θα είναι μόνο δημόσια εθνική συγχρηματοδότηση αυτή, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει και χρήματα από τον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο βέβαια σε τελική ανάλυση κάθε φορά που μιλάμε για δημόσιες συμβάσεις, προφανώς πρέπει να ακολουθούμε τους ισχύοντες κανόνες. Προδοποιούμε βέβαια πάντα τα κράτη-μέλη σχετικά με τις δυσκολίες που υφίστανται και συζητάμε με έναν τρόπο πολύ συγκεκριμένο μαζί τους τι πρέπει να τροποποιηθεί. Προσπαθούμε κατά αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη. Τώρα, το να έχουμε ένα μοντέλο, ένα πρότυπο κοινό για την διάρθρωση των διαφόρων διοικητικών αρχών και δομών είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί επί του παρόντος. Πριν από λίγο στην παρουσίασή μου μίλησα για τη συνεργασία αυτή σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Προσπαθούν ακριβώς να δούνε πώς μπορούν να διαμορφωθούν, να διοργανωθούν οι διοικητικές αρχές των κρατών μελών, ποια προγράμματα κατάρτισης θα μπορούσαν να προβλεφθούν, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των προγραμμάτων. Και έχετε απόλυτα δίκιο όταν λέτε ότι η προπαρασκευαστική φάση των σχεδίων, των έργων είναι πάρα πολύ σημαντική. Κάθε φορά που εξετάζουμε ένα έργο, το οποίο τελικά δεν τα πήγε και τόσο καλά, συνειδητοποιούμε ότι τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στην αρχική του φάση. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο προσπαθούμε ιδίως για τα πολύ μεγάλα σχέδια, έργα, να έχουμε μια υποστήριξη από τον Τζάσπερ και νομίζω ότι εδώ τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά και στα πλαίσια του EIB θα έχουμε και μια πλατφόρμα τεχνικής υποστήριξης Υποστήριξη λοιπόν η οποία προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και βέβαια έχετε όλοι και την τεχνική υποστήριξη η οποία είναι, υπάρχει σε εθνικό επίπεδο και σε ορισμένες χώρες έχουμε βέβαια και τη συμβολή της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ξέρετε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν, πολλές διαφορετικές δυνατότητες προκειμένου να βελτιώσουμε, να διορθώσουμε κάπως το παρασκευαστικό σκέλος, την πρώτη δηλαδή αυτή φάση της κατάρτισης ενός έργου, ώστε να έχουμε καλύτερη προετοιμασία και καλύτερο έλεγχο. Ελπίζω ότι απάντησε στις περισσότερες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Το Μάρτιο θέλω να σας ενημερώσω. Έχουμε μια δημόσια ακρόαση, δεν ξέρω ποιον θα στείλετε από τη Γενική Διεύθυνση. Ε, πάντα πρόσδεκτη θα είναι οι υπάλληλοι που θα στείλετε. Και θα ήθελα εξ ονόματος όλων να σας ευχαριστήσω και πάλι που ήρθατε και ανταλλάξετε απόψεις μαζί σα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ καλό να έχουμε τέτοιες ανταλλαγές απόψεων πάντα. Με χαρά θα παρακολουθήσω, θα, θα διαβιβάσω την ε, πρόσκλησή σας για την επόμενη ακρόαση. Ωραία. Τελειώσαμε λίγο νωρίτερα από ό,τι είχαμε προγραμματίσει την πρωινή μας συνεδρίαση. Διακόπτεται λοιπόν η συνεδρίαση μέχρι τις 3 το απόγευμα. Ευχαριστώ.